Ladies and gentlemen, good morning. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ λάβετε θέσεις γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι αρκετά φορτωμένη η σε διάταξή μας. Και πάλι καλημέρα σας. Σας καλωσορίζω. Για λίγο καιρό, για λίγη ώρα θα ακούτε πολωνικά. Mm. Τη μητρική μου γλώσσα δηλαδή. Θα ήθελα να αναδειχθούν και οι διερμηνείς εδώ. Έχετε λάβει λοιπόν όλη την ημερήσια διάταξη. Εντάξει με τη διερμηνία. Έχετε λάβει, επαναλαμβάνω, την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Όχι, σας ευχαριστώ. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Η γραμματεία σας έχει στείλει και τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης ε, της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας. Πρόκειται για τα πρακτικά της 7ης Ιουλίου του 2014. Αν μέχρι το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης δεν κατατεθούν ε, παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, τα πρακτικά θα θεωρηθούν συγκεκριμένα, χωρίς παρατηρήσεις αμετάβλητα. Παρακαλώ, ε, λάβετε υπόψη ότι έχουμε λάβει την παρέτηση του πρώτου αντιπροέδρου της υποεπιτροπής μας, του κυρίου Γκάλερ, εκπροσώπου του ΕΛΚ. Το ΕΛΚ, η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υπέβαλε την ε, υποψηφιότητα του κυρίου Κρίστιαν Έλλερ για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου της Υποεπιτροπής. Και θα παρακαλούσα τον συντονιστή να μας κάνει την παρουσίαση της υποψηφιότητας. Ευχαριστώ πολύ Ήδη το είχα πει από την περασμένη συνεδρίαση για λόγους τεχνικών ε, αναπροσαρμογών. Αυτό θα ήταν το απλούστερο και ήδη σας έχω ανακοινώσει γραπτός ότι παρετούμε σήμερα και ο συντονιστής του ΕΛΚ προτείνω τον κύριο Δόκτωρ Κρίστιαν Έλαρ ως αντικαταστάτη. Ήδη από την περασμένη θητεία συμμετείχε πάρα πολύ ενεργά στις εργασίες μας ο κύριος Έλερ και θεώρησα ότι ήταν κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση από πλευράς του ΟΕΛΚ. Ε, ε, ο κύριος Κρίστιαν Έλερ είναι μόνιμο μέλος της Υποεπιτροπής ε, Ασφάλειας και Άμυνας και μάλιστα έχει καταθέσει και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων, το Ποθενέσχες. Συμφωνεί δηλαδή με την υποψηφιότητα εσείς συμφωνείτε, υπάρχει συνένεση. Ευχαριστώ. Κύριε, υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι, οπότε θα πρότεινα να εγκρίνουμε την υποψηφιότητα του κυρίου Κρίστιαν Έλερ για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας διαβοήσα με χειροκροτήματα. Παρακαλώ, αν συμφωνείτε. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Έλλερ, ελάτε να λάβετε τη θέση σας στο Προεδρείο. Και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γκάλερ για τη μέχρι τώρα συνεργασία. Ο κύριος Γκάλερ θα παραμείνει μέλος ε, της Επιτροπής και θα είναι συντονιστής του ΕΛΚ. Παρακαλώ κύριε Έλλερ, ελάτε στο Προεδρείο. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να λάβετε υπόψη το διευρυμένο Προεδρείο της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας με βάση το άρθρο 205 του κανονισμού του, Ευρωπαϊκού, του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα η υποεπιτροπή μας να εκχωρήσει οριοθετημένες από τον εσωτερικό κανονισμό αρμοδιότητες στο διευρυμένο Προεδρείο. Γιατί ο φόρτος εργασίας της ε, Επιτροπής καθιστά αναγκαίο για να διευκολύνουμε την κατάσταση, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο διευρυμένο Προεδρείο. Βέβαια εξαιρούνται οι εγκρίσει ε, εκθέσεων, είτε η ίδια πρωτοβουλία ε, τη Υποεπιτροπή Ασφάλεια και Άμυνα, η κατανομή των ακροάσεων, των σεμιναρίων, συγγνώμη, για όλα αυτά τα θέματα θα λαμβάνουν αποφάσει ε, οι συντονιστέ που συμμετέχουν στο Διευρυμένο Προεδρείο. Το Διευρυμένο Προεδρείο θα παρτίζεται από τον Πρόεδρο και του αντιπροεδρου και από του ε, συντονιστέ. Και έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η διαδικασία αυτή είναι σημαντική και η, η έκθεση φυσικά, κάθε έκθεση θα πρέπει να ε, λαμβάνει την έγκριση του Διευρυμένου Προεδρείου της ΑΦΕΤ και να περνάει από τη διάσκεψη των Προέδρων. Συμφωνείτε με την πρόταση αυτή? Δηλαδή να εκχωρήσουμε τέτοιου είδους αρμοδιότητες στο Διευρυμένο Προεδρείο από την Υποεπιτροπή μας. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με τον τρόπο αυτό ακολουθούμε την πρακτική της προηγούμενης ε, κοινοβουλευτικής ε, περίοδου και επομένως πιστεύω ότι πρέπει να διατηρήσουμε την παράδοση και υποστηρίζω την πρόταση αυτή. Εάν δεν υπάρξουν ε, περαιτέρω αντιρρήσεις, εγκρίνεται λοιπόν αυτή η απόφαση και επομένως μπορούμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό στην επόμενη. Θα μπορούμε να κάνουμε τη συνεδρίαση του διευρυμένου Προεδρείου μας που θα λάβει χώρα μετά από την συνεδρίαση της προεπιτροπής μας και στις μεταγενέστερες μας επίσης συνεδριάσεις εγώ θα έχω την ευκαιρία να ανακοινώσω το χρονοδιάγραμμα της επόμενης μας ε, συνεδρίασης. Και τώρα επιτρέψτε μου να περάσω σε δύο πολύ σημαντικά σημεία της ημερησίας διάταξής μας. Καταρχήν να καλωσορίσω θέρμος τον πρέσβη κύριο Μάτσιετ Ποπόφσκι, ο οποίος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Προσκαλέσαμε τον κύριο Ποπόφσκι για να μας ενημερώσει σε σχέση με τα αποτελέσματα της άτυπης συνεδρίασης του, του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών με τη μορφή των Υπουργών Άμυνας που έλαβε χώρα χθες, Τρίτη, στο Μιλάνο. Έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι παρόν ενώπιον της υποεπιτροπής σας. είναι πρόθεσή μου να συνεχίσω να παρίσταμε στις συνεδριάσεις σας εφόσον το επιθυμείτε. Η ενημέρωση αυτή <clears throat> νομίζω γίνεται σε μια σωστή χρονική στιγμή γιατί η συνεδρίαση η άτυπη των Υπουργών Άμυνας έλαβε χώρα χθες. Ήταν μια ιδιαίτερη συνάντηση, πρώτα απ' όλα γιατί ακολούθησε αμέσως την ε, διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία και 22 από τις 28 υπουργούς ήταν πράγματι παρόντες στο Νιούπορτ στη διάσκεψη του ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, το πλαίσιο της συζήτησης επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα τεκτενόμενα στην ε, Ουκρανία, αλλά και στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη, όπως γνωρίζουν όλοι. Ένας τρίτος λόγος για αυτή τη συνάντηση είναι κάπως ε, ειδικού χαρακτήρα, γιατί βρισκόμαστε στα μέσα μιας θεσμικής μετάβασης ε, περιμένοντας την ε, έλευση του νέου ή της νέας ΙΠΑ του εκπροσώπου. Ο κύριος ότι προείδρευσε εξ ονόματος της ΙΠΑ εκπροσώπου, της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Θα έρθω λοιπόν στα επιμέρους θέματα τώρα. Ήταν παρόντες οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ σε αυτή τη συνάντηση. Αυτό είναι πάγια πρακτική και σε αυτή την περίπτωση ήταν ο αναπληρωτής ε, διευθυντής για διοικητής για θέματα ανάλυση ο κ. Κράους και από εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών την Έρβα Λατσού από το τμήμα διατήρησης της ειρήνης που ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της συνάντησης για τις, ε, τους σχηματισμούς μάχης και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Επί της ουσίας, το πρώτο τμήμα της συζήτησης αφορούσε τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου πέρσι αλλά μέσα στα πλαίσια και της κρίσης που των κρίσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα τόξο αστάθειας γύρω από την Ευρώπη που ξεκινά από την Ουκρανία, περνάει από τη Μέση Ανατολή και φτάνει στη Λιβύη και οι Υπουργοί Άμυνας πράγματι εξέφρασαν την ανησυχία τους για αυτή την κατάσταση. Υπάρχει μια διασπορά <clears throat> περαιτέρω συγκρούσεων που πλησιάζουν όλο και περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν εκκλήσεις για μια εντατικοποιημένη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό με το ΝΑΤΟ σε όλες τις ενέργειες που έχουν να κάνουν με τον τομέα της ασφάλειας και άμυνας. Αν δούμε όμως τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2013 για τα αμυντικά θέματα, μπορούμε να πούμε σήμερα ότι τα θέματα άμυνας είναι ακόμα πιο σημαντικά από ό,τι στο παρελθόν υπάρχουν τα έγγραφα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Το ένα είναι ο δικός χάρτης για την εφαρμογή σε σχέση με την, με την πρόταση της Κομισιόν για τον αμυντικό τομέα βιομηχανίας που ενεκρίθη πέρσι τον Ιούνιο και επίσης και η έκθεση προόδου της ΥΠΑ του, του επικεφαλής της υπηρεσίας της ε, εξωτερικής δράσης που διανεμήθηκε πέρσι στον ε, τον πέρσι τον Ιούλιο. Ο κ. Περότσι παρουσίασε επίση το έργο που έχει να κάνει με την εφαρμογή τη ανακοίνωση τη Κομισιόν για τα θέματα αυτά και ακολούθησε και μια σύντομη παρουσίαση τη ε, έκθεση τη Υπάτου εκπροσώπου. Για να τονίσω ορισμένα ειδικά σημεία τώρα. Αυτή τη στιγμή τώρα περατώνουμε τη διαδικασία του πλαισίου πολιτικής για μελλοντική μακροχρόνια αμυντική συνεργασία. Ήταν ένα από τα καθήκοντα που είχε αποδοθεί στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα εύκαμπτο και ελαφρό πλαίσιο θα έλεγα που βασίζεται στην ιδέα ότι μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη διαδικασία συντονισμού, καλύτερο χρονισμό των διαδικασιών, καλύτερα ε, πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ μας. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο αναφέρθηκε είναι το θέμα της χρηματοδότησης των αποστολών και των επιχείρησεων. Παραμένει μια πρόκληση για όλους μας όπως ξέρετε, είτε πρόκειται για πολιτικές είτε πρόκειται για στρατιωτικές αποστολές και ΕΠΑ. Έχουν κατατεθεί μες προτάσεις που είναι υποσυζήτηση από τα κράτη-μέλη. Παραμένει ένα πολύπλοκο θέμα για θεσμικούς, νομικούς και ε, δημοσιονομικούς λόγους. Πρέπει όμως να βρούμε πραγματιστικές λύσεις για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να αντιδρούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και ένα τρίτο θέμα ήταν το θέμα της ταχείας αντίδρασης. Αλλά πέραν μοναχά των σχηματισμών μάχης, τους οποίους θα επανέλθω, η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρουσίασε ένα σύντομο έγγραφο προβληματισμού σε σχέση με την δυνητική χρήση του άρθρου 44 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα επέτρεπε σε μια ομάδα 100 μελών να αναλάβουν μια δραστηριότητα στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ το άρθρο 44, επομένως απλώς εξετάσαμε ορισμένε πρακτικές και νομικές συνέπειες της χρήσης αυτού του άρθρου. Θα συνεχιστεί η συζήτηση, δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη συζήτηση μεταξύ των Υπουργών για το θέμα αυτό αλλά προσδοκούν πολλά κράτη-μέλη ότι η εκπρόσωπο θα μπορέσει να παρουσιάσει και τις απόψεις της για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια, συζητήσαμε τα θέματα των σχηματισμών μάχης. Μετά από την αίτηση πολλών κρατών μελών, που εκφράστηκε στην τελευταία επίσημη συνεδρία των Υπουργών Άμυνα τον ε, Απρίλιο. Εξετάστηκε το θέμα των σχηματισμών. Εδώ το κύριο μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει μια τέλεια κρίση που θα προσαρμόζεται στην έννοια του σχηματισμού. μάχης. αυτό είναι μια έννοια την οποία επεξεργαζόμαστε πολύ καιρό. Δεν θεωρούμε ότι μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Τελικά όμως όλα έχουν να κάνουν με την πολιτική θέληση και η λύση για τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να ξεβρεθεί σε πολιτικό επίπεδο. Ο Υπουργό ε, Άμυνα τη Σουηδία, καθώς και άλλοι υπουργοί, αναγνώρισαν ότι χρειάζεται μια βελτίωση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι παραμένουν σε εμβληματικό ρόλο οι σχηματισμοί μάχης για να δίδονται στρατιωτικού χαρακτήρα απαντήσεις. Τέλος, θέλετε το θέμα και πάλι, όπως είπα, της πολιτικής θέλησης. Ήταν ενδιαφέρον ότι έλαβε το λόγο ο εκπρόσωπο των ΗΕ και ενεθάρρυνε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να χρησιμοποιεί περισσότερο του σχηματισμού μάχη. Πάντα υπεστήριζαν μια τέτοια αντιμετώπιση και η ιδέα των σχηματισμών μάχης είχε αναπτυχθεί μετά από την πρώτη ε, επιχείρηση της Ευρωπαϊκής ένωση το 2003 στην ε, Δημοκρατία του Κονγκό χρησιμοποιώντας τους σχηματισμούς αυτούς. Χθε επίση ξεκινήσαμε μια <clears throat> συζήτηση για τον Ευρωπαϊκό Φορέα ε, Υπηρεσία Άμυνα. Ήταν η δέκατη επέτειος της δημιουργίας της CDA του Ευρωπαϊκού Φορέα Άμυνας. Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα χρονική στιγμή να κάνουμε ένα απολογισμό και μπορούμε να πούμε ότι η υπηρεσία αυτή έχει κάνει θετικό έργο αλλά δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιήσει πλήρως τα κράτη-μέλη την πλήρη δυναμικότητα αυτού του φορέα. Τέλος, υπήρξε και μια συζήτηση σε σχέση με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όσο σκεφτόμαστε τα γεγονότα στην Ουκρανία, Συρία, Ιράκ και Λιβύη, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις άλλες καταστάσεις κρίσης στον κόσμο και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το κέρας της Αφρικής, το Μάλι, η Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, η Βοσνία Ζεγοβίνη. <clears throat> Ήταν λοιπόν για όλα αυτά μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία για τους επικεφαλείς των επιχειρήσεων αυτών να ενημερώσουν τους ε, υπουργούς. Υπήρξαν δύο τμήματα αυτής της συζήτησης. Ένα τμήμα που ήταν οι εκτελεστικές αποστολές Βοσνία, Αταλάντα και Κεντρική Αφρική και επίσης οι αποστολές εκπαίδευσης στο Μαλί και τη Σομαλία και η συμβουλευτική αποστολή στο Κόγκο. Ο στρατηγός ε, Μπάτσελ, ο οποίος είναι επικεφαλής της ε, Αλτέα, τόνισε ότι το προσδοκή της ε, επικείμενες εκλογές στη Βοσνία Ζεγοβίνη και τόνισαν πολλοί υπουργοί ότι βέβαια δεν ήταν ακόμα πρόσφορο από χρονική άποψη να σταματήσει η εντολή της Αλτέα. Πρέπει να ληφθούν επομένως αποφάσεις από το Συμβούλιο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Για την Αταλάντα επίσης υπήρξε σαφής αναγνώριση της επιτυχίας του εγχείρηματο, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπαθίες μας. Έχουν μειωθεί τα επεισόδια πειρατείας από περίπου 170 το 2011 σε δύο μονάχα απόπειρες εφέτος, αλλά φυσικά τα αίτια της πειρατείας προέρχονται από την κατάσταση στην ξηρά στη Σομαλία και υπάρχει συμφωνή μεταξύ των κρατών μελών ότι η αποστολή της Αταλάντα θα πρέπει να παραταθεί μέχρι το τέλος του 2016. Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ΦΟΚΑΡ έχουμε δύο θέματα τα οποία εμπλέκονται. Καταρχήν το θέμα της χρονικής αλληλουχίας. Μέχρι το Δεκέμβριο κανονικά θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η αποστολή, αλλά η, μετά, η μετάδοση τις εξουσίες για τα θέματα αυτά στα Ηνωμένα Έθνη μπορεί να μην λειτουργήσει επαρκώς, γι' αυτό ορισμένοι έχουν ζητήσει να υπάρξει μια παράταση αυτής της αποστολής. Κάποτε θα αποχωρήσει αυτή η αποστολή, αλλά η ανάγκη να εξασφαλιστεί <clears throat> η μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλεια στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι κάτι το οποίο παραμένει ω πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να συζητηθεί το θέμα αυτό. Η συζήτηση αυτή είναι εξελίξη και θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα στην Πολιτική και Στρατιωτική Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε επίση και με τα Ηνωμένα Έθνη. <clears throat> για τις μη εκτελεστικού χαρακτήρα αποστολές εκπαίδευσης και δημιουργίας ικανότητας. Ουσιαστικά υπήρξε ένας απολογισμός. Νομίζω ότι έχουμε κάνει πολύ καλά πράγματα στον τομέα αυτό, ιδίως σε ό,τι αφορά τον αριθμό των στατιών των που έχουν εκπαιδευτεί στο Μαλί και στην Σομαλία. Παραμένουν πολλές προκλήσεις ενώπιών μας, μεταξύ των οποίων η παροχή εξοπλισμού, υπάρχουν πολιτικά και νομικά προσκόμματα για την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού όχι μόνο στρατιωτικού αλλά και εν γέννη, αν θέλουμε να κάνουμε αυτή την εκπαίδευση και να δημιουργήσουμε ικανότητα, το επόμενο επίπεδο θα πρέπει να είναι να διευκολύνουμε την παροχή εξοπλισμού, γιατί αλλιώ αυτοί οι στρατιώτε του οποίου εκπαιδεύουμε δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικοί. Και στι δύο περιπτώσει το Μαλί και τη Σομαλία, τώρα προχωρούμε στο επόμενο επίπεδο προ την παροχή συμβουλών σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση των ένοπλων δυνάμεων του Υπουργείου Άμυνας των χωρών αυτών. Αυτό παραμένει μια πρόκληση, ιδίω για την ε, αποστολή μας στη Σομαλία, η οποία λειτουργεί στο Μογαδίσιο από, το 2000, από την αρχή του 2014 και έχει τώρα πλήρη δύναμη, πλήρη παρουσία. Και τέλος, αναφερθήκαμε και στην αποστολή στο, στη Δημοκρατία του Κονγκό, Προχωρούμε τώρα σε μια μεταβατική φάση, θα μειωθεί η... ο αριθμό των μελών αυτής της αποστολής, θα συνεχίσει όμως το έργο της και θα πρέπει να συμπληρώσει το έργο το οποίο θα επομιστεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στον τομέα των, της μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας. Λοιπόν, αποδίδουν καρπούς οι αποστολές μας, παραμένουν φυσικά προκλήσεις πολιτικού και νομικού χαρακτήρα και φυσικά χρειαζόμαστε διευρυμένους πόρους για να μπορέσουμε να φέρουμε σε πέρα σε αυτό το εγχείρημα σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της τέταρτης γενιάς. Ήταν λοιπόν πυκνές οι συζητήσεις, καταδεικνύουν ότι έχει γίνει για να ενδοθεί συνέχεια στα συμπερασμάτια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2013, αλλά επίσης αντανακλούν και το δύσκολο πλαίσιο το οποίο υπάρχει για τα θέματα ασφαλείας γύρω από την Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρεζοστά για την παρουσίαση. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντονιστές. Αρχής γενομένης από τον κύριο Γκάλερ. Έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποπόφσκι για την ε, παρουσίαση αυτή των πεπραγμένων στην άτυπη σύνοδο. Αναφερθήκατε στο άρθρο 44 που δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί Καταρχήν είναι ένας από τους τομείς που εμείς ανέκαθεν επικρίναμε, ότι δεν αξιοποιούμε ακόμα πλήρως το δυναμικό της συνδίκης της Λισαβόνας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Εσείς έχετε την εντύπωση ότι και δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων που αναφέρετε κι εσείς, κάπως εμφανίζουν κάποια προθυμία τα κράτη-μέλη να το σκεφτούν αυτό, να αξιοποιήσουν πλήρω την πλήρη δυνατότητα που τους δίνει η συνθήκη για δράση. Και για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. είπατε ότι ε, γιόρτασε την ε, δέκατη επέτειο από την ίδρυσή του ε, γενέθλια δηλαδή και πάλι εκεί υποαξιοποιείται το δυναμικό και οι δυνατότητες γιατί δεν το κάνουν αυτό τα κράτη-μέλη τους πεσεύουν τα λεφτά ή δεν θεωρούν ότι μπορούν να συνεργαστούν σε αυτό το τομέα. Και ένα τρίτο που θέλω να ρωτήσω. Αναφερθήκατε στις διάφορες αποστολές και τις επαριθμίσατε. Έχω μια ερώτηση για το Μαλί. Εκεί εκπαιδεύσαμε στρατιώτες. και <laughs> από ό,τι φαίνεται, ο Πρωθυπουργός έχει αναθαρίσει τόσο πολύ που έχει τέτοιο φοβερό στρατό που ε, έκανε μία επιχείρηση ε, για επίδειξης δυνάμεων και για να το πω έτσι, η Μάης τα μούτρα του και σκοτώθηκαν και στρατιώτες ε, τους οποίους εμείς είχαμε εκπαιδεύσει. Είναι πολύ εύθραυστο ακόμα εκεί το κράτος. Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Μήπως χρειάζεται μια παράλληλη προσπάθεια και πολιτικά, όχι μόνο στο στρατιωτικό σχέλος. Ε, μήπως χρειάζεται και πολιτική παροχή συμβουλών εκτός από τη στρατιωτική. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Ο κύριος Πάσκου, ξεραματος των σοσιαλιστών, παρακαλώ. Well. Ευχαριστώ. Εγώ ήρθα να ακούσω βασικά, αλλά το τελευταίο αυτό που είπε ο κύριος Γκάλερ, όταν πήγαμε πριν από δύο-τρία χρόνια και επισκεφτήκαμε τότε στην Ουγγάντα, το κέντρο εκπαίδευσης που τότε ήταν στην Ουγκάντα ε, εμείς ε, απλώς ε, εκπαιδεύαμε το υλικό που βρίσκαμε εκεί και το δυναμικό με αφίβολα αποτελέσματα. Το θέμα δεν είναι μόνο λοιπόν να είναι προετοιμασμένοι και πολιτικά και να τους ενισχύσουμε και πολιτικά. Αν είναι έτσι αρκετά ε, ασταθές το περιβάλλον. Δεν αρκεί πάντα η στρατιωτική εκπαίδευση. Ναι, συμφωνώ, θα πρέπει ίσως να τους εκπαιδεύουμε και πολιτικά, να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε. Και ελπίζω να ληφθούν αυτά υπόψη. Ευχαριστώ κύριε Πάσκου. Ο κύριος Βανόρντεν Εξ ονόματος των συντηρητικών, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως είπε ο κύριος ε, Παπαυσκή και γνωρίζει, οποιαδήποτε συζήτηση για την ΕΠΑΑ ε, φέρνει σε πάρα πολύ δινή θέση το Ηνωμένο Βασίλειο. Από τη μια, δεν θέλουμε να παραμείνουμε αδρανείς και να μην βοηθάμε. Από την άλλη, ε, θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αίσθηση ότι η στρατιωτική παρουσία είναι ε, άχρηστη όσο και αντιπαραγωγική συχνά. Για το άρθρο 44 ε, βάζει και άλλο πρόβλημα και δίλημα. Η ε, επιχείρηση Αταλάντη επέτυχε, λέτε, η λεγόμενη επιτυχία εκεί, η αντιμετώπιση της πειρατείας. Η επιτυχία δεν έχει καμία σχέση με την ίδια την επιχείρηση. Ε, το πιο αποτελεσματικό συστατικό ήταν ότι ε, πάνω στα σκάφη τα ίδια ε, είχαν τη δυνατότητα να προστατευτούν με ενόπλους. Στην αρχή είχαμε μια, ε, ομάδα, ε, μια μονάδα δύναμη ταχείας αντίδρασης 60.000 ε, που αντικαταστάθηκε από τους σχηματισμούς μάχης, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις όπως είναι η Ουκρανία αυτό που χρειαζόμαστε είναι σαφήνεια και ξεκάθαρα μηνύματα που να στέλνουμε σε δεχομένους εχθρούς εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση και να μην δημιουργούμε προβλήματα. Και Προφανώς σε μια κατάσταση τύπου Ουκρανίας αλλά και άλλες καταστάσεις δεν θα πρέπει να ε, ανακοινούμε εμείς εκεί τα πνεύματα και να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Αυτή είναι η ιδέα της ε, ταχείας αντίδρασης ήθελα να αναφέρω και τη συζήτηση στη Ρώμη για μια εχμή του δόρατος ε, τέτοια ομάδα δράσης ε, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. 4.000 και θα εδρεύει στην Πολωνία, αν δεν απατώμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει καθόλου σε αυτό. Για να είμαστε ειλικρινεί, ο μόνος λόγος που θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στρατιωτική παρουσία είναι για να πληρώνει μερικά από τους λογαριασμούς. Γι' αυτό επιμένει η Γαλλία τόσο πολύ. Είναι οικονομικό το κίνητρο. Για να είμαστε ειλικρινεί, σε αυτό το τομέα έχουμε εκτελέσει, πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σενάρτα από τους Φιλελεύθερου. Ευχαριστώ. Η Ευρώπη, να κάνουμε ένα παραλληλισμό, φαίνεται να είναι τεράστια στο μάχη με ένα μικρό κεφάλι. Αυτή είναι μια λυπηρή πραγματικότητα και θα μας φέρει σε μια μακροχρόνια συζήτηση για να προσπαθήσουμε να εντάξουμε κάτι που υπάρχει στην Ευρώπη που είναι μια εξωτερική, κοινή εξωτερική πολιτική και μια ε, ε πολιτική άμυνας που θα πρέπει να είναι πραγματική και όχι απλώς θεωρητική. Η μάχη με ομάδες, τα battle groups με τις 1500 στρατιώτες είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν μπορεί να ε, παρά να περιοριστεί σε συγκεκριμένε ε, μικρή εμβέλεια ε, στρατιωτικέ επιχειρήσει. Δεν μπορεί να επεκταθεί σε πολλέ επιχειρήσει αυτό ο σχηματισμό των μάχημων μονάδων. Επίση, έχουμε την πρόταση για την, ε, ε το σχηματισμό τη δύναμη ταχεία αντίδραση, ώστε να γίνουμε πραγματικό φορέα εξωτερική πολιτική και όχι απλώ να πληρώνουμε λογαριασμού. Μιλήσαμε τώρα για την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση στο Μαλί. Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Στο Μαλί ε, ιτήθηκαν οι φουνταμεταλιστές και το αρέκι και Μόρας χάρη στο, στο αίμα που έχησε ο στρατός του Τσάντ. Ε, εκεί έδρασε επί τόπου ο στρατός του Τσάντ. Και ε, συνέβαλε και ο Γαλλικός στρατός με, με βομβαρδισμούς, γιατί δεν έδωσε το παρόν εκεί ο στρατός του Μαλή. Και ακόμη και όταν έδρασε ήταν παταγώδηση η αποτυχία του. Ας μην είμαστε λοιπόν ε, πολύ συγκαταβατική και επίκης με τους εαυτούς μας. Είναι σημαντικός, ε, η σημαντική εκπαίδευση, αλλά η συντήρηση είναι ακόμη πιο σημαντική, διατήρηση, γιατί αν δεν δώσουμε στην τοπική κυβέρνηση τους πόρους για να κρατήσει τη διαδικασία αυτή, τότε ε, το θέμα θα είναι μόνο μισθολογικό. Το θέμα είναι ποιος θα μείνει με τα χρήματα. Και τελικά δεν θα έχουμε καμία ουσιαστική πρόοδο. Αυτό ισχύει και για τη Σομαλία. Και εκεί, όπως στην Ουγγάντα, είχαμε εκπαίδευση σομαλικών τμήματων που μερικές φορές εντάχθηκαν στις μονάδες της ΣΑΜΠΑΧ. Το θέμα είναι όχι πόσους εκπαιδεύσαμε, αλλά τι αποτελεσματικότητα έχει το σώμα που δημιουργήσαμε και τι παρουσία επιτόπου στο πεδίο της μάχης. Και κάτι που είπαν και είναι αλήθεια, το θέμα είναι ποιος επιλέγει στους ε, σχηματισμούς, γιατί θα πρέπει να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη, στην πραγματικότητα. Γιατί οι τοπικές κυβερνήσεις που μερικές, φορέ είναι απλώς ε, φιλές, φιλετικές κυβερνήσεις, ουσιαστικά θέλουν τη δική τους φιλή και με, το, με την ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δημιουργούν σχηματισμούς για να τους εξυπηρετούν. Είναι θέμα λοιπόν διαφθοράς. Ουσιαστικά χρησιμοποιούνται μερικέ φορέ από φυλέ τέτοιες, σχηματισμοί και επιτόπου πολλέ φορέ διαλύονται γιατί δεν υπάρχουν χρήματα και τα χρήματα αυτά τα έχουν καρποθεί οι φύλαρχοι για τους δικούς τους σκοπούς. Τι εχέγγυα έχουμε για την αποτελεσματικότητα αυτών των μονάδων, ώστε πραγματικά να μπορέσουν και οι κυβερνήσεις για να, διαχειρίσουν, να διαχειριστούν αυτές τις μονάδες που εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει και εκπαιδεύσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νάρτ. Η κυρία Λέζινγκ τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ε, Ευχαριστώ πολύ τις ερωτήσεις του κυρίου Γκάλερ και των άλλων συναδέλφων για την υποστήριξη τη στρατιωτική σε ασταθή κράτη. Θέλω να την υποστηρίξω πάρα πολύ ρητά. Είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ και έχει να κάνει και με πωλήσει όπλων σε διάφορες περιφέρειες. Κοιτάξτε στη Συρία τι γίνεται, στο Ιράκ. Κανείς δεν ξέρει πού φτάνουν τελικά αυτά τα όπλα, σε ποια χέρια πέφτουν και τελικά ποιες ε, ε, μονάδες ένοπλες υποστηρίζονται από στρατιώτες που εμείς εκπαιδεύουμε. Ε, τώρα όμως θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, ε, σε δύο τομείς. Πρώτον, τι γίνεται με το μηχανισμό ε, Αθηνά, στο άρθρο 41, παράγραφος 2, ε, ορίζονται οι στρατιωτικές δαπάνες και οι αμυντικές δαπάνες και απαγορεύονται και δεν ε, υπάρχει αυτή τη δυνατότητα, η δυνατότητα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό να χρηματοδοτούν χρηματοδοτούνται στρατιωτικές και αμυντικές δράσεις. Ε, ο μηχανισμός των Αθηνών όμως έχει υποστεί κάποια αναδιάρθρωση και δεν είναι δυνατόν να καταβάλλονται κατά αποκοπή ποσά ε, για ε, αμυντικούς σκοπούς. Είναι παράνομο αυτό. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει μια επιφύλαξη του Κοινοβουλίου και ε, διαιρωτώ με πώς μπορεί αυτή να είναι δεδομένη όταν δίνουμε έτσι γενικά κατά αποκοπή ποσά σε στρατιωτικές δράσεις. Και ρωτώ, το έχετε συζητήσει με τους Γερμανούς και πώς σκοπεύουν να ξεπεράσουν αυτό το σκόπελο του Κοινοβουλίου. Και επίσης η μονάδα ταχείας επέμβασης. Ε, εδώ είναι ένα πάγιο αίτημα στην Επιτροπή να υπάρχει ε, μια τέτοια δυνατότητα που να μπορεί να αναπτύσσεται μέσα σε δύο έως πέντε ημέρες. Μα πώς μπορεί να περάσει μέσα από ένα κρατικό κοινοβούλιο μια τέτοια απόφαση, αν πρόκειται για δύο με πέντε μέρες. Σας ρωτώ, εκεί που συναντήσετε εκπροσώπους των κρατών μελών, τα συζητήσατε αυτά, τα έθεσαν εκείνοι υπόψη σας και πώς απαντάτε. Και ποιες στρατηγικές έχετε ε, προτείνει και ευχαριστώ. Τσαμπάιας για τους Πρασίνους. Κυρία Τσαμπάιας. Ε, σας, παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας γιατί μιλάω σουηδικά. Ε, υπάρχει το θέμα της χρήσης των ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρξει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί για τη χρήση αυτών των αεροσκαφών. Και εδώ θα πρέπει να ε, υπησέλθει ο Ευρωπαϊκός Αμυντικός Φορέας. Επίσης, το burden sharing, η κατανομή του άχτους, υπήρξε αυτό αντικείμενο συζήτησης. Και επίσης, οι προϋπολογισμοί άμυνας. Ξέρω ότι οι χώρες της Ευρώπης σε πολλές περιπτώσεις έχουν μειώσει τους προϋπολογισμούς τους για την άμυνα, ενώ το ΝΑΤΟ έχει ζητήσει να γίνει το αντίθετο, να υπάρξει αύξηση των προϋπολογισμών. Τι θα γίνει με τα θέματα αυτά. και επίσης η δημιουργία αυτών των σχηματισμών μάχης σημαίνει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να υπομισθούν ένα μεγαλύτερο κόστος από ότι στο παρελθόν. Επίση, η παράδοση φρεγάτας Μιστράλ στη Ρωσία είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει. Εγώ είδα με βάση τις ε, ειδήσει που έχω παρακολουθήσει μέχρι τώρα ότι το θέμα αυτό δεν έχει ακόμα επιληθεί πλήρως. Επίση το θέμα τη ενέργεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει. Δεν είναι μονάχα όμω το θέμα τη ενέργεια και τη ε, τροφοδοσία με ενέργειε. Και επίσης, πρέπει επίση να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των αποβλήτων που δημιουργούνται με την ευρωπαϊκή πολιτική ενέργεια και πώ θα αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη τα θέματα αυτά. Thank you, madam. Uh, I would like to ask it... Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος ε, ε, του FDD θέλει προ το λόγο. Όχι. Ο κύριο Έλερ τώρα. Mr. Ambassador, I would like to ask you... Um, Θα ήθελα να, να σας ρωτήσω, κύριε Πρέσβη, δύο ε, ε πράγματα. Παρά ε, τα όσα είπε ο Τζέφρι Όρντενς, για τον άτο και το σεβασμό που πρέπει να τρέφουμε. Ε, μα και οι δύο ε, ε, οργανισμοί έχουν την ίδια μέρημνα για το πρόβλημα των αερομεταφορών. δεν έχουμε λύσει το στρατηγικό μας πρόβλημα, ένα ενδιάμεσο. και στάδιο έχουμε για ένα κοινό μηχανισμό ΝΑΤΟ και σχηματισμό μάχης. Ε, σε ποιο βαθμό είναι αυτό πραγματικά επιχειρησιακό και ε, πώς θα γίνει αυτή η κοινή ε, δράση. έχω και μια ερώτηση για τα στρατηγία. Ουσιαστικά οι δομές του ΝΑΤΟ και πρακτικά αναπερίπτωση αναλαμβάνουν αυτή τη διοίκηση όταν τα χρησιμοποιούμε ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ε, το παράδειγμα, μια επέμβαση της Τουρκίας ας πούμε να αποτρέψει τη χρήση αυτών των σχηματισμών. Και έχω και μια ερώτηση για τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό μιλήσατε για μια, την επαιτειακή αυτή συνεδρίαση. Ωραία, αλλά είναι και επέτειος των προβλημάτων, ε, όχι μόνο της ε, ίδρυσης του οργανισμού. Τι γίνεται με τη χρηματοδότησή του. Τώρα αρχίζουμε τη συζητήση για τον προπολογισμό του 2015 και οι εξηγήσει που ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά ήταν κάπως χλιαρές το Κοινοβούλιο αποφασίζει για κάποιο μηχανισμό ενδεχομένως από την πρόταση ορίζον 2020, δηλαδή τεχνικά είναι εφικτό αυτό, αλλά στην πράξη δεν έχουμε βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση που να ξέρουμε ξεκάθαρα ποια θα είναι η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Αυτό το έχετε σκεφτεί, σας έχει προβληματίσει και το θέμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού, πού θα μπορούσαμε να βρούμε τα χρήματα και με ποιο μηχανισμό να ε, τα διοχετεύουμε σε έργα του ΕΝΤΑ. Ευχαριστώ. Περιμένουμε τον κύριο Τζέμς Απατουράη, που είναι αναπληρωτής βοηθός Γενικού Γραμματέα ε, και το πρόγραμμά μας είναι πολύ φορτωμένο. Θα ήθελα να θέρμα παρακαλέσω τους ε, ομιλητές μας να είναι λακωνικοί. Ο κύριος Στέτινα είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, έχω μία ερώτηση που με απασχολεί και προσωπικά. Πριν από ένα περίπου μήνα πήγα στην Ανατολική Ουκρανία και είδα με τα μάτια μου ένα, εν, μία μονάδα εθελοντών που δεν έχουν κανένα εξοπλισμό. Με... Δεν έχουν ούτε καλά όπλα, δεν έχουν καν αλεξίσφαιρα γυλαίκα, δεν έχουν καν αρβίλες. Μάχονται με κανονικά παπούτσια. Ίσως λοιπόν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κάπως ε, το Ουκρανικό στρατό. Το επόμενο σημείο της ημερήσης διάταξης, κύριε Στέτιν, αφορά την Ουκρανία. Μήπως ε, θα θέλετε να περιμένετε λίγο και να θέσετε την ερώτηση αργότερα. Ναι, δίκιο. Έχετε καλύτερα αργότερα. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ποπόφσκι, θα ήθελα να σας θέσω το εξή ερώτημα. Εν ώψη της κρίσης που αντιμετωπίζουμε στην Ουκρανία, τι διδάγματα <clears throat> μπορούμε να αντλήσουμε, τι συστάσεις, τι προτάσεις προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Φορέα ή τι ζητήθηκε από τον ε, Αμυντικό Φορέα να προτείνει για να εξασφαλίσουμε ότι πράγματι θα είμαστε έτοιμοι μέσα στα πλαίσια της ε, ΚΕΠΑ αλλά και του ΝΑΤΟ να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες οι οποίες θα προκύψουν σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα των εξοπλισμών μας, τον καλύτερο την καλύτερη εκπαίδευση των ε, στρατιωτικών δυνάμεών μας και τις άλλες ανάγκες οι οποίες μπορεί να προκύψουν. Σε αμυντικό επίπεδο. Να σας ρωτήσω επίσης κατά πόσο το Συμβούλιο έχει διαμορφώσει κάποιο μηχανισμό αξιολόγησης των επιπτώσεων των κυρώσεων που θα επιβληθούν σε ό,τι αφορά την ε, προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού από την πλευρά της Ρωσίας και ιδίως σε ό,τι αφορά τα αγαθά δυτής τεχνολογίας και τη δυνατότητα κάποιες τρίτες χώρες να παράσχουν στη Ρωσία εξοπλισμό που εμείς θέλουμε να εμποδίσουμε να φτάσει ως εκεί. Για το Ιράκ και τη Σύρια. Είχαμε την κυρία Ιβάσκοβα στην Επιτροπή μας, η οποία τόνισε ιδιαίτερα ότι οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί που δίδουν τα κράτη-μέλη μας στις ε, στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράκ και πιο συγκεκριμένα στους Πεσμεργά, στις δυνάμεις του, της κουρδικής συνιστώσεως του Ιράκ εναντίον της ε, του Ισλαμικού κράτους, ουσιαστικά είναι ανεξέλεγκτες αυτές οι παραδόσεις όπλων. Δεν, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς φτάνει εκεί. Τι θα κάνει λοιπόν το Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας. Και είπα τι εκπρόσωπος για να τεθεί κάποια τάξη και να υπάρξει κάποιο συντανισμό σε αυτές τις προσπάθειες και επίσης να εξασφαλιστεί μια συνέργεια μεταξύ των προσπαθειών που γίνονται και σε επίπεδο εσωτερικών και ασφάλειας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των λεγόμενων ξένων τσίχαδιστών που προέρχονται από την Ευρώπη. Για τη Λιβύη επίσης. Η Λιβύη είναι ένα Αφγανιστάν κοντύτερα στην Ευρώπη. Είπατε ότι η Λιβύη ήταν στο μυαλό όλων, αλλά η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που δεν είναι θέμα του να είναι απλώς το πνεύμα μας. Είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με χειροπιαστό τρόπο να κάνουμε κάτι. Σε ποιο βαθμό εμείς συντονίζουμε τις προσπάθειές μας μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις αραβικές χώρες που είναι όμορες της Λιβύης για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που είναι τόσο σοβαρή που θα τη χαρακτήριζα πραγματικά σαν ένα Αφγανιστάν στο κατόφλι μας. Και επίσης να σας ρωτήσω κατά πόσο έχει εξεταστεί η κρίση του ιού έμπολα, όχι σαν θέμα ασφάλειας, αλλά σαν μια δυνητική ε, χημική ή βιολο... απειλή χημικού ή βιολογικού πολέμου και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μιλήσατε επίσης και για τα θαλάσσια θέματα, την θαλάσσια διάσταση της ΚΕΠΑ. Είπατε ότι η Αταλάντα θεωρείται μια επιτυχία. Μα ξέρουμε πόσες πράξεις πειρατείας έγιναν στον κόλπο της Γουινέας στην Αφρική και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εκεί γιατί υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά σκάφη τα οποία έχουν εμπλακεί σε ενέργειες οργανωμένου εγκλήματος με την ε, λαθρεμπορία κλεμμένου πετρελαίου από, το, από την περιοχή της Νιγηρίας και επίσης για το πλαίσιο κυβερνοάμυνας υπάρχουν κάποιες ε, συνέπειες που προέκυψαν ενώπιση των κρίσεων με τη Ρωσία και την Ουκρανία για να αναθεωρήσουμε αυτό το πλαίσιο για την κυβερνοάμυνα. Και τέλος να πω ότι βρίσκω πραγματικά αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι ενώπιον όλων αυτών των κρίσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τα κράτη-μέλη μας δεν μπορούν να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία για να υπάρξει μια αναθεώρηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της και σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γόμες. Τρεις ομιλητές μας έχουν απομείνει στον κατάλογο και θα ήθελα να τον ολοκληρώσω. Ο κύριος Ζέμκε. Έχετε το λόγο κύριε Ευρωβουλευτά. Εδώ βρισκόμαστε ακόμη στο πρώτο σημείο της, της συνεδρίασης και αυτό θα περιοριστώ σε αυτό το πρώτο σημείο. Θα ήθελα να σας θέσω συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχήν, ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Είπατε ότι εορτάστηκε η δέκατη επέτειο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Θα πρέπει τώρα να κάνουμε έναν απολογισμό της αποτελεσματικότητας του οργανισμού αυτού. Ερωτώ λοιπόν, πώς ε, κρίνεται την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Γιατί εγώ έχω πολλές αφιβολίες ως προς το κατά πόσο είναι αποτελεσματικός αυτός ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνα Προσπάθησα να σας παρακολουθήσω προσεκτικά και αν δεν κάνω λάθος μιλήσετε και το Αφγανιστάν. Τι σημαίνει αυτό. Ε, αν το ΝΑΤΟ αλλάξει φέτος τη φιλοσοφία, θα αλλάξει φέτος τη φιλοσοφία του και απέναντι στο Αφγανιστάν ή ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει μία ανάληψη δράση γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόιτ. Καλημέρα σας, κυρία Πρόεδρε. Εξοχότατε. Διατέλεσα δημοσιογράφος εγώ στην προηγούμενη ζωή μου και θα ήθελα να ε, συνεχίσω ε, εκεί που σταμάτησε η Άννα εδώ παρακαθήμενη, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις το απαιτούν. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση στο Ιράκ και στη Συρία έχει επιδεινωθεί σφόδρα. Και αφού του έφυγαν από το Ιράκ οι συμμαχικές δυνάμεις, η χώρα διαλύεται όλο και περισσότερο. Μεγάλες περιοχές ε, στο Ιράκ δεν είναι πια στα χέρια της κυβέρνησης και στον έλεγχό της και έχουν πέσει στα χέρια αυτών που αυτό αποκαλούμε Ισλαμικό κράτος, ε, παρόλο που δεν είναι ούτε Ισλαμικό ούτε κράτος, τρομοκράτες είναι. Πρόσφατα ε, είχαμε αυτούς τους αποτρόπαιους θανάτους δολοφονίες των Αμερικανών και ο πρόεδρος Ομπάμα χθε το βράδυ ανακοίνασε στο Λευκό Οίκο ότι και στη Συρία ε, θα επιτεθούν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, στο Ισλαμικό κράτος, στο Ιράκ και στο Λεβάντε. Για πρώτη φορά και επιμένει και προς τους συμμάχους του ο Ομπάμα να ε, καταπολεμήσουν αυτό το Ισλαμικό κράτος. Ε, χιλιάδες όμως ε, ξένοι μαχητές και από τα κράτη-μέλη μας πολεμούν στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους και μπορεί να αποτελέσουν και κίνδυνο για τις ίδιες τους χώρες και τους πολίτες της. Πώς σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει σε αυτό που ζήτησε ο Ομπάμα, μια ευρεία συμμαχία. Ποιος θα απαντήσει σε αυτή την έκκληση του Ομπάμα από την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούχνερ. Meine Frage richtet sich... Η ερώτησή μου απευθύνεται ε, στη χρήση των μη επαδρομένων αεροσκαφών, όπως ε, ε, λέει το πρόγραμμα. Τι προβλέπετε. Θα είναι μόνο αναγνωριστικά αυτά. Αυτές οι πτήσεις θα είναι μόνο αναγνωριστικές. Πώς έχει η δομή της διοίκησης εκεί. να μην υπάρξει αμελής χρήση σε ένα θέατρο πολέμου. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ήδη σήμερα στις σειράξεις υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου χρειάζονται στρατιωτικές αναγνωριστικές πτήσεις με μη επανδρομένα ε, αεροσκάφη. Τα ευρωπαϊκά αυτά αεροσκάφη πώς θα ε, χρησιμοποιούνται και ποιος αποφασίζει για τις πτήσεις αυτές ε, για να δώσει τη διαταγή. Κύριε Πρεζευτά, σας δίνω το λόγο και σας θα παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ε, ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό και μακροσκελής ο κατάλογος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία. Και θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω και κάποιες ερωτήσεις για να μην επαναλαμβάνομαι. Για τη χρήση του άρθρου 44. Για το κατά πόσο υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία για τη χρήση του τώρα. Ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε συμπέρασμα, γιατί μερικές χώρες είναι υπέρ της ε, ε, αξιοποίησης το έπακρο του δυναμικού της συνθήκης της Λισαβόνας και το άρθρο 44 δεν είναι, ε, δεν ισοδυναμεί με την μόνιμη συνεργασία. Είναι διαφορετική η διατύπωση. Οπότε κατοχυρώνεται η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωση Χρησιμοποιείται σε διαφορετική κατάσταση. Πάντως θα συνεχιστεί η συζήτηση σε πιο τεχνικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν πολλά πολιτικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα που θα πρέπει να συζητηθούν. Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και κατά πόσο αξιοποιείται στο έπακρο το δυναμικό του. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός είναι οργανισμός άμυνας και ασχολείται με αμυντικά σχέδια, που είναι μακρόπνοα γιατί χρειάζεται πολύς χρόνος για να αποδώσουν καρπούς αυτά τα προγράμματα. Είναι πολύ χρονοβόρα. Και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας δημιούργησε ήδη αυτό το περιβάλλον της καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας αλλά και με την αμυντική βιομηχανία. Και βλέπετε ότι στις συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας έχουμε όλο και μεγαλύτερη παρουσία της αμυντικής βιομηχανίας και υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον και ετοιμότητα για δέσμευση, αλλά δεν είναι εύκολο να ποσοτοκοποιήσουμε αυτό το ενδιαφέρον. Γιατί και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Άμυνας έχει οικονομικά προβλήματα εξαιτία τη συρρήκνωση προϋπολογισμού και έχουμε δύσκολε συζητήσει με αμεληταία ποσά στον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπω είπε ο κύριο Σέλερ, χρειάζονται κάποιε συνέργειε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επανέλαβε και ε, είναι ερώτηση στο Μιλάνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει τι προπαρασκευαστικέ δράσει για συγκεκριμένα σχέδια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα. Πέρυσι το είχε αναγγείλει, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο και φαντάζομαι θα το αναλάβει αυτό και η Νέα Επιτροπή και θα το προωθήσει γρήγορα. Γιατί αυτό ενδιαφέρει και την αμυντική βιομηχανία και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην αμυντική βιομηχανία. Και Έχουμε βέβαια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις ε, στο ΚΕΠΑ που δεν, ε, προ... δεν χρηματοδοτούνται από υπολογισμό του ορίζοντα 2020. Αλλά είναι και αυτό ένα σημείο στο οποίο θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο το συντομότερο δυνατό. Για την κατάσταση στο Μαλί. Είναι αρκετά εύθραυστη κατάσταση στο Μαλί. Και όπως είπε ο κύριος Γκάλερ ότι οι στρατιώτες που, που εκπαιδεύσαμε εμείς πήγαν, στη, ε, πήγαν στο βορρά και απέτυχαν, δεν φταίνε εκείνοι. Ε, αυτοί που έδωσαν, έφταγαν αυτοί που έδωσαν τις διαταγές. Και πραγματικά διδαχθήκαμε από τα παθήματά μας και τελικά διαπιστώσαμε ότι δεν έφταγε η εκπαίδευση που προσφέραμε. Αλλά αν δεν χρησιμοποιούνται σωστά οι πόροι, και δεν είναι σωστέ ε, οι εντολέ που δίνονται, η ήττα είναι αναπόφευκτη. Και νομίζω ότι τα κατάλαβαν αυτό και οι θύνοντε στο Μαλί. Και εμείς παρέχουμε και στρατηγικές συμβουλές και συνεχίζουμε και την εκπαίδευση των στρατιωτών. Και πρόκειται και το πέμπτο τάγμα του στρατού του Μαλή να εκπαιδεύσουμε τώρα. Σε ό,τι αφορά την πειρατεία, προσπαθώ να συγκεντρώσω τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν για την πειρατεία. Ο κύριος Βανόρντεν είπε ότι ε, η επιτυχία της Αταλάντης οφείλεται στην παρουσία ενόπλων στα σκάφη. Εν μέρη ναι, αλλά Ακριβώς η παρουσία ενόπλων στα σκάφη ήταν τμήμα της επιχείρησης Αταλάντη. Δεν ήταν ξεχωριστή δραστηριότητα. Και φυσικά αντλούμε και διδάγματα από την επιχείρηση Αταλάντη και στα πλαίσια του, της ε, Διεθνούς Ομάδας Επαφής για την ε, πειρατεία στις ακτές της Σομαλίας. Και μάλιστα εμείς έχουμε την Προεδρία φέτος, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα δούμε κατά πόσο αυτά τα διδάγματα μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και σε άλλες περιπτώσεις όπως τον κόλπο της Γουινέας. Μπορεί να ακούγονται αφηρημένα όλα αυτά, αλλά πραγματικά τα διδάγματα αυτά που συγκεντρώνουμε θα τα συμπιλήσουμε ε, σε μια διεθνή μελέτη και θα τα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε πού μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αλλού. Επίσης, η χρήση ιδιωτικών επιχειρήσεων ασφάλειας ε, για την ασφάλεια των πλοίων, ο τρόπος επικοινωνίας, για παράδειγμα, που θα ενεργοποιούνται και οι μονάδες του ΝΑΤΟ σε συγκεκριμένες περιοχές. Και, επαναλαμβάνω, αυτό που κάνουμε στο κέρας Αφρικής μπορούμε να το κάνουμε και στον κόλπο της Γουινέας. Για τις μάχημες μονάδες τώρα και τη δύναμη ταχές αντίδρασης. Είναι αποφάσεις του ΝΑΤΟ για την δύναμη ταχεία αντίδραση που είναι αιχμητοδόρατο και αναφέρθηκε στο Μιλάνο στη συνεδρίαση, αλλά δεν συζητήθηκε εκτενώ. Είναι απόφαση του ΝΑΤΟ. Και κάνουμε κάποιε συγκρίσει με τι αποφάσει του ΝΑΤΟ για θέματα ταχεία αντίδραση. Και η συνεργασία με το ΝΑΤΟ είναι πολύ εύχριστη και πρακτική και έχει βελτιωθεί αισθητά του τελευταίου μήνε. Και βοήθησε και σε αυτό βέβαια την επιτάχυνση της συνεργασίας η κρίση της Ουκρανία. Αλλά φυσικά δεν έχουμε ε, ρόλο εμείς στην ανάπτυξη της δύναμης του ΝΑΤΟ και της δύναμης ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Και ο γενεσιουργός της λόγος είναι διαφορετικός. Ιδέεται με, το άρθρο 5, ενώ οι μάχημες ομάδες ε, εντάσσονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Τώρα, ε, για τη χρηματοδότηση και την αναθεώρηση του μηχανισμού της Αθηνάς που θα ξεκινήσει εντός ολίγου. Τα ερωτήματα βέβαια είναι τα ίδια. Θα μπορέσουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της κοινή χρηματοδότησης. Αυτό κυρίως σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των στρατευμάτων. Το θέμα αυτό ανήκει στην, στον διακυβερνητικό τομέα. Δεν έχουμε κοινοτική συμβολή και κανένας δεν το πρότεινε. Δεν υπάρχει τέτοια ιδέα. Θα δούμε που θα φτάσουμε. Η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2011 αλλά θα αντιλήσουμε ε, διδάγματα και από την ανάπτυξη στην κεντροαφρικανική δημοκρατία που ήταν ε, σχετικά αργή. Πάντως ε, ελπίζω τα κράτη-μέλη να δείξουν μεγαλύτερη προθυμία για ανάμειξη στη συζήτηση αυτή. Ο ρόλος των κοινοβουλίων σε ό,τι αφορά την έγκριση των αναπτύξεων. Δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη αυτές τις μάχημες ομάδες, τα battle groups και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης τέτοιων μάχημων σχηματισμών είναι πιο αργά σε σχέση με την ανάπτυξη της δύναμης ταχύς αντιδράσης του ΝΑΤΟ. Για τις στρατηγικές μεταφορές δεν σχεδιάζουμε κοινοτική συμβολή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτό θα συζητηθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης του μηχανισμού της Αθηνάς. Πάντως, αυτό που είναι ενδιαφέρον και επιτυχές είναι η μονάδα μας στο Eindhoven που είναι συντονιστική για τις μεταφορές που λειτουργεί πολύ καλά και, χρησιμοποιείται και χρησιμοποιήθηκε και στην ανάπτυξη στην κεντροαφρικανική δημοκρατία αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Για τα μη επαδρομένα αεροσκάφη, τα drones, αυτό που συζητήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα drones είναι οι τεχνικές προδιαγραφές και πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ευρωπαϊκή τεχνολογία. Δεν μιλούμε για ευρωπαϊκό στρατηγείο ή για ε, δικής μας ε, ιδιοκτησίας drones, για ευρωπαϊκά ε, μη επαδρομένα αεροσκάφη. Είναι θέμα περισσότερο τεχνικά και όχι λήψη αποφάσεων ποια είναι η αλυσίδα λήψης αποφάσεων και εντολών. Αυτό δίνεται σε εθνικό επίπεδο και δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Τώρα για τους αλλοδαπούς διχαντιστές και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε. και θα επιληφθούν και οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, παρόλο που και εμείς παρακολουθούμε εκ του στο ζήτημα. Τώρα, είναι πρόσφατη η έκκληση για ένα νέο συνασπισμό για το Ιράκ, πρόταση του, των Ηνωμένων Πολιτειών στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μια έκκληση που απευθύνθηκε προς συγκεκριμένα κράτη-μέλη, προς μεμονωμένα κράτη-μέλη και όχι προς ε, οργανώσεις. Και θα δούμε στην πράξη πώς θα υλοποιηθεί αυτό. Και τέλος, δύο ακόμη θέματα καταρχήν ε, αμυντικές, ε, προμήθειες στον αμυντικό τομέα και η επίπτωση των κυρώσεων σε πωλήσει αμυντικού εξοπλισμού προς τη Ρωσία. Όλα αυτά ε, συνεχίζονται να εξετάζονται και στις 11 θα συνεχίσει τη συζήτηση Κορεπέρ, θα γίνουν περαιτέρω περιορισμοί. Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, φυσικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό, αλλά έχουμε, είχαμε διαβήματα με προσπολές πολλές τρίτες χώρες που έχουν επαφές εμπορικές με τη Ρωσία να μην προχωρήσουν την παράδοση αμυντικού εξοπλισμού. Και τέλος, για το Αφγανιστάν. Δεν έχουμε ξεχάσει το Αφγανιστάν. Ο πρόεδρος Βαν Ρομπόι μίλησε στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ για το Αφγανιστάν, στην συγκεκριμένη συνεδρίαση που αφιερώθηκε στο θέμα αυτό και μίλησε για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποστολές εκπαίδευση αστυνομικών, με μεταρρύθμιση του αστυνομικού σώματος. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή συμμετοχή και συνεχίζουμε να ενεργοποιούμαστε στο Αφγανιστάν και μάλιστα αφιερώσαμε, αφιερώνουμε 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Σήμερα, ναι, παρακαλώ κύριε, κύριε Νάρτ. Κύριε Πρέσβη, δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να πω ότι όταν είναι κάτι το οποίο είναι ουσιώδες θα πρέπει να τύχει απάντησης. Η αποτελεσματικότητα των μονάδων που εκπαιδεύουμε όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικό αλλά σε επίπεδο δράσεις στην πραγματικότητα. Τόνισα την αδυναμία της αλυσίδας διοίκηση. Έχω μεγάλη εμπειρία για τα θέματα του πολέμου στην, άμυν, στην ε, έρημο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε εύκαμπτες ε, ομάδες οι οποίες να διευθύνονται από λοχαγούς ή υπολοχαγούς από, ατό, από άτομα τα οποία έχουν πραγματική ικανότητα, όχι να υπάρχει αδυναμία στην αλυσίδα διοίκησης. Πέραν του να κάνετε μονάδες στα χαρτιά να δημιουργείται μονάδα στα χαρτιά. Τι εγγύηση έχουμε ότι είναι πραγματικά αποτελεσματικά τα στελέχη αυτών των μονάδων και ότι διατηρούνται και δεν διαλύονται αυτές οι μονάδες όταν δεν υπάρχει πληρωμή για τους στρατιώτες ή γιατί έχουν φιλετική βάση ούτως ή άλλως από την αρχή. Μπορείτε να απαντήσετε εν συντομία κύριε Ποπόσκη και μετά και έχω κλείσει φυσικά τον κατάλογο των αγορητών. Ναι, να σας πω το εξής. Γνωρίζουμε το πρόβλημα αυτό το οποίο αναφέρατε και γι' αυτό ιδιαίτερα στο Μαλί κάνουμε επανεκπαίδευση των ε, δυνάμεων οι οποίες αποστέλλονται στο βόρειο τμήμα του Μαλί. Όταν γυρίζουν χρησιμοποιούμε τα διδάγματα τα οποία έχουμε αποκομίσει από την ανάπτυξή τους και επανεκπαιδεύονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την εθνοτική φιλετική σύνθεση αυτών των μονάδων παραμένει ένα θέμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει μια στρατηγική συμμετοχή και από την πλευρά των κυβερνητικών αρχών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν οι κυβερνήσει ότι τα εθνικά στρατεύματα έχουν μια πιο εξισορροπημένη σύνθεση μετά από τον πόλεμο. Ακριβώ μετά από τον πόλεμο ήταν καθαρά σε φιλετική βάση και εκεί έχετε δίκιο. Πρέπει να τροποποιηθεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η πρόεδρο. Κλείνουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτού του σημείου στην ημερησία διάταξή μα. Και επανερχόμαστε εννέα μήνες σχεδόν ακριβώς μετά την εκκίνηση της ε, απόφασης που ελήφθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2013 και είμαστε και εννέα μήνες περίπου πριν από το Συμβούλιο του Ιουνίου του 2015 που θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο σε βάθος για τα θέματα αυτά, τα αμυντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ακούσει λοιπόν σημαντικά θέματα να αναφέρονται κατά τη διάρκεια, να τη διάρκεια αυτής της συζήτησης και περιλαμβάνεται και στην έκθεση που θα συζητήσουμε στο επίπεδο του διευρυμένου μας Προεδρείου αργότερα. Σας ευχαριστώ. Κάνουμε μια διακοπή ενός λεπτού και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης.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 Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν παρακαλώ κάντε το ησύχος και ηρέμος και ταχαίως κυρίως. Επαναλαμβάνουμε τη συνεδρίασή μας. Παρακαλώ καθίστε Καθίστε λοιπόν. Να καλωσορίσω δύο μιλητές. οι οποίοι θα λάβουν το λόγο στο επόμενο σημείο της ημερήσια διαταξής μα, και θα αναφερθούν στις προκλήσεις οι οποίες προκύπτουν από την κρίση στην Ουκρανία την ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις ένοπλες επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα εκεί. Χαιρετίζω λοιπόν τον αναπληρωτή βοηθό Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ κύριο, κύριο James Απατουράη που είναι ο πρώτος μας ομιλητής και ο οποίος θα μας παρουσιάσει την οπτική γωνία του ΝΑΤΟ για την κρίση αυτή. Και ο επόμενο ομιλητής μας είναι πιο γνωστός, είναι ο πρέσβη Ματσέη Ποπόσκι, ο οποίος είχε την καλοσύνη να συμμετάσχει και στην προηγούμενη μας συζήτηση σε σχέση με το άτυπο συνέδριο Συμβούλιο <clears throat> Υπουργών Άμυνα. Κύριε Απατουρά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε έχω αρχίσει να γνωρίζω λίγο καλύτερα αυτή την αίθουσα και αυτή την επιτροπή. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να με παρών ενώπιόν σα. και δίνει και στον ΝΑΤΟ ελπίδα όταν μπούμε στο νέο κτίριό μας σε κάποιο ομιχλώδες ε, μέλλον γιατί βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει ένα ωραίο κτίριο όπως το δικό σας. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα το οποίο μου θέσατε ε, για να λάβω το λόγο μαζί με τον φίλο μου το Ματσιέ είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά κυριάρχησε στη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ πριν από λίγε μέρες και υπάρχουν πολλά ε, στοιχεία αυτή τη συνδιάσκεψης που μπορεί να ενδιαφέρουν τους συναδέλφους. Μία πτυχή της κρίσης της Ουκρανίας είναι φυσικά η σχέση του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία. Εν συντομία, αυτό το οποίο προέκυψε από την διάσκεψη του της Ουαλίας είναι ότι δεν έχει αλλάξει η σχέση μας με τη Ρωσία, αλλά έχει παγώσει ουσιαστικά η πρακτική συνεργασία. Έχουμε την ευκαιρία για πολιτικό διάλογο, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής και να σας πω ότι δεν είναι ιδιαίτερα καρποφόρος αυτή τη στιγμή αυτός ο πολιτικός διάλογος. Δεν είχαμε λοιπόν μεγάλη πρόοδο για τα θέματα αυτά. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στην Ουαλία τόνισαν ότι ο στόχος μας θα πρέπει να είναι μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία Πρέπει όμως να είναι μια εταιρική σχέση με μια Ρωσία η οποία με σταθερό και συνεχτικό τρόπο σέβεται το διεθνές δίκαιο και τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Και αυτά δεν είναι μονάχα γενικόλογα σχόλια. Υπάρχει μια δέσμευση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν η Ουκρανία αποφάσισε να παραδώσει τα πυρηνικά της όπλα, στην Βουδαπέστη υπήρξε η ανάληψη υποχρεώσεων από τη Ρωσία να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Ρωσίας, της Ουκρανίας, συγγνώμη, και φυσικά τώρα έχει παραβιάσει ουσιαστικά την ε, ανεξαρτησία της ε, Ουκρανίας με την παρουσία σταθευμάτων, την υποστήριξη σε αποσυστικές τάσεις, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά. Δεν πρόκειται λοιπόν μονάχα για μια παραβίαση σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Είναι ένα θέμα πολύ μεγάλης ανησυχίας για όλη την Ευρώπη ότι η Ρωσία έχει ε, ουσιαστικά παραβιάσει τόσο σημαντικές υποχρεώσεις και άλλες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει της τελικής πράξης του Ελσίνκη. Ανοίγω τώρα μια παρένθεση. Ε, αυτό δεν ε, δίνει διαβεβαιώσεις σε χώρες όπως η Βόρεια Κορέα ή το Ιράν ότι αν ε, καταστρέψουν τα πυρηνικά τους όπλα ή τα αποσύρουν θα εξασφαλίζεται η ασφαλειά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα της εμπιστοσύνης που έχει χαθεί μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη ότι η Ρωσία μπορεί να λειτουργήσει μέσα στο σύστημα που έχει εξασφαλίσει την ασφάλεια στην Ευρώπη για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι η Ρωσία έχει τη διάθεση να λειτουργήσει μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να έχουμε μια προβλέψιμη σχέση με τη Ρωσία αν η Ρωσία θέλει να αναθεωρήσει αυτό το σύστημα το οποίο έχει λειτουργήσει και να εφαρμόσει τη θέλησή της στους γειτονές της. Αυτό δεν είναι μονάχα κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Άμα δείτε την νομοθεσία της Ρωσίας, τη ρητορική της Ρωσίας, τις θέσεις της Ρωσίας από τότε που ανέλαβε την εξουσία ο κ. Πουτίν, είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα. Η Ρωσία δίνει το δυνα... το... τη δυνατότητα στον εαυτό της να επιβάλλει τη θέλησή της ακόμα και στρατιωτικά εκεί που υπάρχουν ρωσόφωνοι, πολίτες με ρωσικά διαβατήρια ή και βάσει πιο ασαφών κριτηρίων που αφορούν τη ρωσική παρουσία μπορεί να φτάνουν μέχρι την Αλάσκα λοιπόν τα ρωσικά συμφέροντα ή μέχρι και τις χώρες μας. Ξεκινά λοιπόν μια πάρα πολύ δύσκολη και επεπλεγμένη σχέση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και διάβασα σήμερα ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει αναλάβει απόλυτη, ε, απόλυτα την εξουσία στον τομέα της ε, στρατιωτικής βιομηχανίας της Ρωσίας. Έχουν ήδη δοκιμάσει ένα, πύραυλο πυρηνικού, ένα πυρηνικό πύραυλο στη Ρωσία. Πρέπει λοιπόν τώρα να κατανοήσουμε ότι οι σύμμαχοι μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ δεν θεωρούν ότι η Ουκρανία είναι μεμονωμένη περίπτωση και όταν σταματήσουν οι εχθροπραξίες δεν θα γυρίσουν τα πράγματα σε μια φυσιολογική κατάσταση όπως ελπίζουμε. Είδαμε Γεωργία, τη Γεωργία, την Μολδαβία, τώρα την Ουκρανία να υπάρχει μια στάση της ε, Ρωσίας η οποία εφαρμόζει μια πολιτική η οποία είναι αποσταθεροποιητική για την Ευρώπη. Θα επιζητήσουμε λοιπόν μια σταθερή σχέση, μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι η Ρωσία επιζητεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον πρέπει να σκεφτούμε για τις σχέσεις μας με την Ουκρανία. Είδατε τις ανακοινώσεις που έχουν προέλθει από την Ουκρανία. Υπάρχει ιδιαίτερη ε, αλληλεγγύη και από τη δική μας πλευρά για την Ουκρανία και την εδαφική ακεραιότητά της. Έχουμε εγκρίνει μια σειρά από σχέδια που θα βοηθήσουν την Ουκρανία για την μακροχρόνια ανάπτυξή της στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από την πλευρά του ΝΑΤΟ εξοπλίσει το ΝΑΤΟ την Ουκρανία για να ε, αντιμετωπίσει τα θέματα ασφαλεία της. Δεν θα το κάνει αυτό το ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε όμως και θα κάνουμε μέσα από τα σχέδια αυτά είναι να βοηθήσουμε την Ουκρανία να έχει καλύτερες δομές διοίκησης και άμυνας, επιμελητίας, κυβανοάμυνας, τυποποίησης των εξοπλισμών της, στρατηγικές επικοινωνίες, πώς να μπορέσει να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τις αμυντικές της ικανότητες. Αυτό δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλουμε να βοηθήσουμε όμως και την Ουκρανία να διαχειριστεί καλύτερα <clears throat> τα θέματα ε, θεραπείας και περίθαλψης των στρατιωτών της που έχουν τραυματιστεί και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ελπίζοντας ότι χάρη στη δική μας συμβολή και τη συμβολή των ε, συμμάχων μας, θα μπορέσει να υπάρξει αποκλιμάκωση και πέρα των εχθροπαξιών, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια τελική λύση η οποία σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της ε, Ουκρανίας. Αυτό είναι απαράγραπτο για μας. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε χωρίς να κλιμακώσουμε περισσότερο την κρίση για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντιμετωπίσει και να επιλύσει αυτή την κρίση. Ένα τρίτο σημείο, και τώρα περνάω προς τα δυτικά, της Ουκρανίας, τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τις χώρες οι οποίες υφίστανται πίεση από τη Ρωσία να μεταστρέψουν την, την πορεία τους, μάλλον τις χώρες προς τα Ανατολικά, η Γεωργία, η Μολδαβία και άλλες χώρες, που είναι υποπίεση από τη Ρωσία. Έχουμε δημιουργήσει ένα πακέτο υποστήριξης προς τη Γεωργία που θα επιτρέψει τη Γεωργία να βελτιώσει τις αμυντικές της ε, ικανότητες, να εργαστεί περισσότερο για την ε, ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν και στην περίπτωση της, ε, της Μολδαβίας να ενισχύσουμε την αμυντική τους ικανότητα. Δεν θέλουν να γίνουν τμήμα του ΝΑΤΟ, αλλά θέλουμε να τους βοηθήσουμε να είναι σε θέση να διαπιλέξουν τη δική τους γεωπολιτική στρατηγική. Ως ΝΑΤΟ δεν θέλουμε να αναγκάσουμε κάποια χώρα να διαλέξει ή τη Δύση ή την Ανατολή. Αν η Ουκρανία αλλάξει την πολιτική της και ξέρετε το έκανε η Ουκρανία μέχρι το 2008 ήθελε να είναι μέλος του ΝΑΤΟ, τώρα έχει περάσει σε μια στάση περισσότερο αδέσμευτη της χώρας σε ό,τι αφορά τους στρατιωτικούς σχηματισμούς. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Ουκρανία χωρίς να επιβάλλουμε κάποια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αντισταθούν στις πιέσεις της Ρωσίας που θέλει να τις υποχρεώσει να αποστραφούν από την Δύση οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά. Ένα τέταρτο στοιχείο και δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό που προήλθε από τη διασκέψη κορυφή μα. Είναι σαφέ ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ασφάλεια για του συμμάχου μα από το ΝΑΤΟ. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία έχει επενδύσει σημαντικά σε αμυντικές ικανότητες, σε στρατιωτικές ικανότητες. Έχει αυξήσει μέσα σε πέντε χρόνια κατά 50% τον αμυντικό της προϋπολογισμό, 750 δισεκατομμύρια αμερικανικά δολάρια θα επενδύσει τα επόμενα 6 χρόνια σε εξυγχρονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων και μόνο. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι αφού εξυγχρονίσουν τις δυνατότητές τους μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και είναι έτοιμες να τις χρησιμοποιήσουμε. Επίσης υπάρχει το λεγόμενο υβριδικό μοντέλο όπως είδαμε στην Ουκρανία μια, ένα μείγμα στρατιωτικών και πολιτικών εργαλείων ενέργειες πληροφόρησης και αποπληροφόρησης, διείσδυση σε πολιτικό χώρο, κυβερνοεπιθέσεις, χρήση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού ή πρώην στρατιωτικών, συσσόρευση στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας. Όλα αυτά είναι ένα, ένα πλέγμα το οποίο χρησιμοποιεί η Ρωσία και το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε προχωρήσει σε δύο ενέργειες. Καταρχήν πρέπει να δώσουμε διαβεβαιώσει τους συμμάχους μας στα ανατολικά και αυτό με τη χρήση μικρών, τονίζω, μικρών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία, τις τρεις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, ώστε να μπορεί να υπάρξει υποδοχή μεγάλων, μεγαλύτερων στρατιωτικών δυνάμεων αν χρειαστεί. Δεν δημιουργούμε <clears throat> μάχημες μονάδες εκεί, αλλά κέντρα υποδοχής εάν χρειαστεί για να μπορέσουν να υποδεχθούν στρατιωτικές δυνάμεις και αυτό έχει να κάνει με την ιδιαίτερη ε, επαγρύπνηση και την ικανότητα ταχεία αντίδραση να μπορούμε μέσα σε 48 ώρες να μεταφέρουμε στα θέματα τα οποία θα γίνουν θα τύχουν υποδοχή από αυτούς τους σχηματισμού. Εκεί θα τους υποδέχονται και θα μπορούν να αναπτύσσονται μέσα σε 48 ώρες και τα υπόλοιπα ακολουθούν ω επιμελητία. Ε, διαβεβαίωση, ανασυγκρότηση ε, γιατί υπάρχει αυτή η νέα ανησυχία σε, προς Ανατολάς. Ε, και πολύ σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν για τον προϋπολογισμό. Ε, συμφώνησαν όλοι οι σύμμαχοι να σταματήσουν τη μείωση του προϋπολογισμού και να προσπαθήσουν να αφιερώσουν το 2% του ΑΕΠ μέσα σε 10 χρόνια στις αμυντικές δαπάνες. Αυτός είναι ο στόχος. Να δούμε αν θα φτάσουμε εκεί. Ακούμε κάποια εθαρρυντικά πάντως μέχρι τότε. Και ε, το 5 και το 6 το ανέφερα μαζί. Ε, σας είπα, η κρίση στην Ουκρανία κυριάρχησε πάρα πολύ στη Σύνοδο Κορυφής ως θέμα και ε, αναθεωρήσαμε την ευρωπαϊκή ασφάλεια και το ρόλο που καλείται να παίξει το ΝΑΤΟ εκεί. Και ένα τελευταίο, ένα από τα συμπεράσματα ήταν ακριβώς με το υβριδικό μοντέλο, Χρειάζεται πολύ πιο στενή συνεργασία μεταξύ των διεθνών οργανισμών. Μπορεί το ΝΑΤΟ να αναλάβει τα στρατιωτικά, αλλά όταν υπάρχει υβριδική απειλή, χρειάζονται και άλλα στοιχεία τα οποία ανέφερα. Θα πρέπει να ενσωματωθούν στην απόκριση που θα δοθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξει. Σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων και επιτελείων έχουμε πολύ καλή συνεργασία και στο μέλλον φαντάζομαι ακόμα καλύτερη. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Ε, απατουράει. Τώρα θα δώσω και λίγο χρόνο στον πρέσβη, κύριο Ποπόφσκι. Και μετά από μια πολύ ε, ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Παρακαλώ να μας δώσετε τώρα την ευρωπαϊκή προοπτική και ε, διάσταση ε, της κρίσης στην Ουκρανία και πώς προτίθεται να δράσει ή ήδη δρά η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι συμφωνούμε απολύτως τη δέσμευση αυτή προς την ε, εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στην προσέγγιση δεν υπάρχει παραμικρή διαφορά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Τώρα βέβαια τα συμπεράσματα που εξάγουμε εμείς μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικά λόγω και της ε, διαφορετικής εντολής που έχει ο κάθε οργανισμός. Εγώ θα απαντήσω ε, πόσο επηρεάζει η κρίση της Ουκρανίας την ΚΕΠΑ και την ΕΠΑ. Ε, θέλω να το χωρίσω σε δύο σκέλη, το πρόθεσμο και ε, μέσο πρόθεσμο πρώτα και μετά κάποια πιο μακροπρόθεσμα στοιχεία. Όταν κοιτάμε πόσο χρόνο και ενέργεια αφιερώνουμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Ουκρανία, θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά κυριαρχεί η κρίση αυτή αυτόν τον καιρό. Συνεχίζεται η συζήτηση για τις κυρώσεις. Έχουν ληφθεί αποφάσεις, πλην όμως δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί και οι συζητήσεις μεταξύ κρατών μελών συνεχίζονται σήμερα, ε, την ώρα που μιλάμε και αργότερα. Προωθούμε τη Συμφωνία Σύνδεσης και το Κοινοβούλιο έχει να παίξει το ρόλο του την άλλη εβδομάδα ε, και για μια πιο στενή εμπορική συνεργασία και ελπίζω ε, η Βουλή της Ουκρανίας η Ράντα να ε, κυρώσει όπως έχει σχεδιαστεί. Θα βοηθήσουμε την Ουκρανία να προετοιμάσει τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου και επίσης ε, βεβαίω εξακολουθούμε να ανισχούμε και να αγωνιούμε για την οικονομική κατάσταση. Γιατί όσο είναι τόσο έφραυστη η οικονομία, πράγμα που συμβαίνει, δεν μπορούμε να μιλούμε για μια σταθερότητα πιο μακροπρόθεσμη της χώρας. Άρα χρειάζεται και μακροοικονομική αρρωγή και βοήθεια και όπως ξέρετε έχει δημιουργηθεί δική ομάδα ε, Task Force στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δημιουργία ικανοτήτων που ανέφερε ο James. Ε, ε, συμφωνούμε και έχουμε ένα επιμερισμό εργασίας ξέρουμε πολύ καλά ποιος έχει επιφορτιστεί με τι. Σε επίπεδο πρέσβεων ε, είχαμε συχνά ε, συνεδριάσεις όταν ε, υπάρχει το στρατιωτικό σκέλος και παροχή συμβουλών είναι θέμα του ΝΑΤΟ και δεν μπαίνουμε σε αυτά τα χωράφια ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στην πολιτική δημιουργία ικανοτήτων. Υπάρχουν ήδη κάποια προγράμματα εκεί και τρέχουν που δεν χρειάζεται να τα επανεφεύρουμε και αυτά είναι έργα που έχουν να κάνουν με τον εισαγγελέα, επί παραδείγματι, ε, και τώρα ασχολούμαστε με τις ε, ε, αρχές επιβολής του νόμου, αστυνομία, είναι μια αποστολή συμβουλευτική η UIN στην Ουκρανία. Νομίζω είναι 57 η συμβουλή οι οποίοι μεταβαίνουν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός και ε, είναι συμβουλευτική, επαναλαμβάνω, δεν έχει καθόλου εκτελεστική δράση. Μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα αρχίζουν να λειτουργούν οι αρχές Οκτωβρίου. Και σε πλήρη συνεργασία και διαφάνεια πάντα. Υπάρχει μια φυσική ε, συμπροματικότητα πάρα πολύ θετική με τον ΝΑΤΟ. Τώρα, πιο συστηματικά και μακροπρόθεσμα με συνέπειες για την Ένωση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, την ΕΠΑ. Είπε ο Τζέιμς πόσο δραματική είναι αυτή η υπόθεση ε, για την ακαιρεότητα των οργανισμών ασφαλείας είτε είναι ο ΑΣΕ, ε, το, ε, τα Ηνωμένα Έθνη, η Συμφωνία για τον Αφοπλισμό, η συνθήκη αυτή, ε, πιέζονται πάρα πολύ και απειλούνται από τα όσα συμβαίνουν. Παραδόξως, η κρίση που προκάλεσε η Ρωσία ενίσχυσε και αναζωγόνησε τη διατλαντική κοινότητα. Αν δείτε τη διακήρυξη που ενέκρινε η Σύνοδος Κορυφής, πρόκειται για μια νέα προσέγγιση, ραπροσμό ε, του Ατλαντικού. Έχουμε συσφίξει πλέον τις σχέσεις και έχουμε και την πρόθεση να διατηρηθεί αυτή η στενή ε, συνεργασία ε, ακέραιη. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασφάλεια χρειάζεται επανεξέταση. Πράγμα που συμβαίνει. Ε, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Θα επηρεάσει σίγουρα και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και λειτουργεί η επόμενη ε, τη εκπρόσωπος, ε, από την οποία ζητήθηκε, όπως θυμάστε, το Δεκέμβριο ε, να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική. Πριν την κρίση, το Δεκέμβριο, πριν ξεσπάσει η κρίση. Και είπα ότι εκπρόσωπος έχει την εντολή να παρουσιάσει την ανάλυση της στο Συμβούλιο εντός του 2015. αριθμητικό στόχο δεν έχουμε για τις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη, αλλά αντιλαμβανόμαστε, και αυτό φάνηκε πάρα πολύ και από πολλές παρεμβάσεις υπουργών στο τελευταίο άτυπο Συμβούλιο υπέθα ε, στο Μιλάνο, ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά ε, τις δεσμεύσει τους για την ασφάλεια και την άμυνα. Είτε είναι σύμμαχοί του ΝΑΤΟ είτε όχι. Θα πρέπει πραγματικά να γίνει αυτό έτσι με έναν τρόπο συντονισμένο και σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Επίσης θα πρέπει να το ανακοινώνουμε και στον κόσμο να το επικοινωνούμε αυτό. Ο κόσμος έχει συνηθίσει ότι η ασφάλεια και η ειρήνη είναι κάτι το δεδομένο. Καμία σχέση δεν είναι τώρα ε, συμβατικός ο πόλεμος, καμιά φορά είναι υβριδικές ε, αυτές οι καταστάσεις σχεδόν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κατόφλι μας. Και ποιες είναι οι συνέπειες. Θα πρέπει να είμαστε στο ύψος των περιστάσεων και να απαντήσουμε στις εκκλήσεις που γίνονται επανειλημμένα και στις κρούσεις από την άλλη πλευρά του ε, Ατλαντικού Ακούσαμε ε, την ε, ομιλία του Υπουργού Γκέιτς. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Και δεν έχει σημασία αν θα χρησιμοποιηθούν υπό τη σημαία του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Εθνική, στο βαθμό που υπάρχουν. Ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. το είπε και ο Τζέιμς. Αυτή η κρίση επέδρασε πολύ θετικά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΝΑΤΟ αν δείτε ε, το ανακοινοθέν της Συνόδου Κορυφής που είναι και μακροσκελές και πάρα πολύ πυκνό από την Ουαλία, ποτέ δεν είδα τόσο πολλές αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε κανένα έγγραφο του ΝΑΤΟ. Πράγμα πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ ε, δεν είναι μόνο θεσμός προς θεσμό, αλλά είναι και γενικότερα για την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο, στο, ε, στο Σαχέλ, πολέμηση πειρατείας και ένα ε, πλήθος άλλων ζητημάτων. Στη συνεργασία με λοιπόν και το πνεύμα που μας διέπει για την συμπληρωματικότητα, έρχεται αυτό να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει ε, την φυσική κατανομή αρμοδιοτήτων. Επιστρέφει το ΝΑΤΟ στο βασικό του ρόλο άρθρο 5, ε, αποτροπή ε, παρουσίας σε μαχικό έδαφος και βεβαίως θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσήλωσή μας και σε άλλα θέατρα μαχών και την ε, συνεργασία μας με άλλους φορείς που δεν μπορούν από μόνοι τους να δράσουν, είτε είναι το ΝΑΤΟ είτε είναι ο ΙΕ. Για να ολοκληρώσω, η κρίση στην Ουκρανία σίγουρα θέτει ένα νέο πλαίσιο τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013. Είναι πραγματικά επίγουση η κατάσταση και θα πρέπει να ε, δείξουμε σοβαρότητα στις δεσμεύσεις μας για θέματα ασφάλειας και άμυνας και αυτό θα είναι προς όφελος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά και του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ποπόφσκι. Σας ευχαριστούμε κυρία Πατουράη. Και πριν δώσω το λόγο στα μέλη της υποεπιτροπής μας, στους λοιπούς ευρωβουλευτές, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη της Ουκρανίας, τον κύριο Κωνσταντίν Γελισέιεφ σε μια κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίαση του διευρυμένου Προεδρείου της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Εκεί οι πολιτικές ομάδες, ε, τα μέλη και εκπρόσωποι της ε, Υποεπιτροπής μας ε, ενημερώθηκαν για την ουκρανική προοπτική και τις απόψεις της ουκρανικής κυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Θα ήθελα να αλλάξουμε λίγο το διαδικασία, γιατί η κυρία Καηλή, που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, για τη σχέση με την Ουκρανία, έχει πολύ λίγο χρόνο και μπορεί πολύ λίγο χρόνο να είναι μαζί μας, γι' αυτό μου ζήτησε να πάρει πρώτη το λόγο. Έχετε το λόγο κυρία Καηλή. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στη συνεδρίαση και να σας ε, ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας. Ε, γιατί ε, κλιμακώθηκε η κατάσταση ε, χωρίς να και αγνώντας την δική μας δέσμευση για άμυνα. Γνωρίζω ότι ο ρόλος του ΝΑΤΟ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και έχουν ξεκινήσει νέες συζητήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε γιατί δεν είμαστε πιστικοί ως ΝΑΤΟ. Ποιες είναι οι νέες ε, στρατηγικές δεσμεύσεις ε, που θα πρέπει να αναλάβουμε, γιατί στην Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας ε, επικεντρωθήκαμε σε περισσότερα θέματα τακτικής και φυσικά χρειαζόμαστε ένα σχέδιο δράσης ετοιμότητας και πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο σχέδιο δράσης, αλλά ποια είναι η βασική στρατηγική για την κλιμάκωση. Περισσότερες κυρώσεις, αυστηρότερες κυρώσεις ή μόνο αυτό το σχέδιο δράσης ετοιμότητας. Ποια είναι η γνώμη σας. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας τη συνεργασία και μεταξύ μας, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, αλλά και με τη Ρωσία και να δείξουμε με σαφήνεια τα σύνορά μας και τις κόκκινε γραμμές μας. Και επίση να ενισχύσουμε την, το πρόγραμμα ασφάλεια, περιλαμβάνοντας και τα θέματα ενέργειας, σταθερότητα και επίση ελαστικότητα ό,τι αφορά την αντίδραση στην κρίση στα πλαίσια τη Ευρωατλαντική συμμαχία. Όπως είπατε, το ΝΑΤΟ αναφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής πολύ πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν. Πιστεύετε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε περισσότερο ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και να συμβάλλουμε περισσότερο σε μια καλύτερη αντίληψη περί ασφάλειας και πιο ολιστική και σφαιρική. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα μακροσκελέστατο κατάλογο μιλητών. Θα ήθελα να ολοκληρώσω τώρα τον κατάλογο. Θα σας το διαβάσω Πρώτα όμως θα δώσω το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Πρώτα ο κύριος Γκάλερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θα μιλήσω γερμανικά. Θα ήθελα να πω το εξή και να το τονίσω. Δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση στην Ευρώπη μεταξύ κρατών και μέσα σε κράτη μέσα στην Ευρώπη που να δικαιολογεί τη χρήση βίας και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Ρωσία με ένα τρόπο ο οποίος είναι απειρχαιωμένος προσπαθεί να ασκήσει πολιτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τύχει της κατάλληλης απάντησης. Λυπάμαι για το γεγονός ότι η Ρωσία επέλεξε αυτή την οδό, αλλά έχουμε το δικαίωμα και το καθήκον να προστατεύσουμε τον τρόπο ζωής μας, την δημοκρατική μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι λοιπόν η βασική αρχή την οποία θέλω να τονίσω και κατά τα άλλα εγώ θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου με τα συμπεράσματα του ΝΑΤΟ ιδίω τις ε, εκ νέου διαβεβαίωσης που δόθηκαν στους ε, ανατολικούς μας συμμάχους και εταίρους. Πιστεύω ότι όλα αυτά υπήρξαν ναι. θετικά στο παρελθόν. Θέλαμε να ενισχύσουμε και την ε, σχέση μας μεταξύ των δύο οχθέων του Ατλαντικού. Αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει σε πολύ περισσότερες ε, δυνατότητες να αυξήσουμε και τη δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης από την πλευρά μας και στα πλαίσια της κρίσης Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, αλλά σίγουρα αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει και σε βάθος όπως μας έχει υποχρεώσει να το κάνουμε η ρωσική πολιτική. Δυστυχώς. Και λόγω της κρίσης αυτής θέλω να έρθω στο εξή ερώτημα πόσο σοβαρά λαμβάνουμε υπόψη το στόχο του 2% σε ό,τι αφορά την, ε, τις δαπάνες εξοπλισμού. Έχει εξεταστεί αυτό από την αρμόδια επιτροπή της ΕΝΤΑ του Αμυντικού Φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουν αποδεχτεί οι Υπουργοί Άμυνας πέραν των αφηρημένων δηλώσεων υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα ληφθούν, γιατί εγώ θυμάμαι το στόχο του 0,7 στην αναπτυξιακή πολιτική, ο οποίος είχε τονιστεί ρητορικά, αλλά δεν είχε εφαρμοστεί καθόλου στην πράξη. Ελπίζω τα πράγματα θα είναι καλύτερα εδώ. Μία ακόμα ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν το ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις επίσημες δηλώσεις των Ρώσων. Θυμάμαι το λόγο του κύριου Γερασίμοφ το Ιανουάριο του 2013, όπου ουσιαστικά περιέγραψε αυτό το οποίο γίνεται σήμερα στην Ουκρανία. Και αυτός ο λόγος ήταν διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου του, στα ρωσικά φυσικά, αλλά πώς είναι δυνατόν το ΝΑΤΟ να μην έχει λάβει γνώση αυτής της δήλωσης και να μην έχει αντιδράσει σε μια τέτοια δήλωση. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε. Σας ευχαριστώ. Θέλω να ζητήσω τώρα από τα μέλη της Επιτροπής μας να είναι ιδιαίτερα σύντομη στις παρεμβάσεις τους, γιατί έχουμε ένα πολύ μακροσκελή κατάλογο μιλτών και ο πρέσβης Ποπόφσκι θα πρέπει να φύγει σύντομα, επομένως θα πρέπει να του δώσουμε και τη δυνατότητα να απαντήσει στο τέλος των παρεμβάσεών μας. Ο κύριος Πάσκο τώρα, εξ ονομάτως Σοσιαλιστικής Ομάδος. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι γνωρίζετε ότι όταν αυτά ξεκίνησαν η βασική σκέψη που είχα ήταν πόσο δίκιο είχαμε στην αρχή του 90 που ζητήσαμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Τότε ορισμένοι έλεγαν ότι καλά υπάρχουν ε, εγγυήσει, ε, ακόμα και τώρα βρήκα δημοσιεύματα που λένε ότι ήταν σφάλμα να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Καθόλου σφάλμα δεν ήταν. Με τη διαφορά ότι τότε θεωρήσαμε ότι η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ θα έστελνε τα σωστά μηνύματα σε ενδεχόμενους αντιπάλους και κυρίως για επιστροφή της Ρωσίας. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό και γι' αυτό χρειάζεται στρατηγική επαναβεβαίωση, ε, πράγμα που ελήφθη. Ένα δεύτερο. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Πούτιν δρά και με όρους πολιτικούς, όσο και στρατιωτικούς. Ακριβώς έχει μια υβριδική έτσι, προσέγγιση και σχέση ε, στρατιωτικών και διπλωματικών ε, δραστηριοτήτων και άλλων ενεργειών. Διότι έχει πραγματικά ένα στρατηγικό στόχο που προσπαθεί να εφαρμόσει με τακτικά μέτρα έτσι ώστε να αποφύγει μια στρατηγική απάντηση σε αυτό. Οπότε, για παράδειγμα, αν κοιτάξετε την κατάπαυση του πυρός που ήταν ακριβώς την εβδομάδα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και ήρθαν νέες κυρώσεις και είδαμε ότι ακριβώς εκείνη την εβδομάδα συνέβη και αυτό. Και τι επέτυχε, αναβολή της επιβολής των κυρώσεων. αλλά ευτυχώ δεν κατάφερε να αναμειχθεί στι αποφάσει του ΝΑΤΟ να επηρεάσει. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο και έρχομαι να ρωτήσω εγώ. Έχουμε επίγνωση του γεγονότος ότι ε, κάτω από το ραντάρ για να αποτρέψουν τη δράση μας. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στο ανακοινωθέν που το καταδεικνύουν αυτό. Μια ευέλικτη απάντηση από το το χρειάζεται ε, και ταυτόχρονα ό,τι και να κάνουμε, κάθε κίνησή μας έχει, πώς να το πω, δύο στόχους. Πρώτον, να στείλουμε ένα μήνυμα αποτροπής και να κάνουμε τον κύριο Πούτιν να σταματήσει και σε περίπτωση που συνεχίσει να είμαστε σε θέση να αμυνθούμε. Αλλά φαίνεται ότι αυτά δεν αποτρέπουν τον κύριο Πούτιν. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο θα έλεγα, όπου εμείς κάπως έχουμε δεμένα τα χέρια μας, διότι δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη. Δεν τον αποτρέπουνε. Και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας ε, ε, αίσθηση, αν έχει επίγνωση των άτων όλων αυτών. Και προς τον κύριο Ποπόφσκι. Επιτέλους ξυπνήσαμε στην ε, Ευρώπη, στην άμυνα. Τόσες φορές εδώ έχουμε συζητήσει τις προσδοκίες μας από το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου και τώρα μόλις αρχίζει η αφύπνιση και ανακαλύψαμε ότι Α, μάλιστα, τώρα το κατάλαβαν οι φίλοι μας, τι μας περιβάλλει. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τι να κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πάσκο. Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς τους ομιλητές να είναι λακωνικοί. Και στους συντονιστές και στους υπόλοιπους ομιλητές. Αλλιώς ε, θα χρειαστεί να ενεργοποιήσω το χρονόμετρο και να σας κόβω. Ο κύριος Σνάρτ. εκ μέρους των φιλελευθέρων. παρακαλώ. Χρόνο φίδο. Ανάλογα με το μέγεθος και των πολιτικών ομάδων. Θα προσπαθήσω. Η Ουκρανία είναι η τρίτη φάση μετά το Κωσυφοπαίδιο, την Απχαζία και την Οσετία. Το πρόβλημα ήταν ο κατακαιρματισμός της συμφωνίας ε, για το Κόσοβο και ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη αυτή. Και το ΝΑΤΟ ξεπέρασε την εντολή του στην περίπτωση της Λιβύης. Παρόλο που ε, και εγώ είμαι πεπισμένος για την αναγκαιότητα ανατροπής ε, του Καντάφη. Αναμφισβήτητο αυτό. Αλλά έχουμε μια κλιμάκωση. Και έχουμε... Ε, παρουσιάζουν ως σχεδόν ε, μια διαδικασία Συγγνώμη, ε, ξέρω λίγα Ισπανικά, αλλά δεν έχουμε μετάφραση, διερμηνία από τα Ισπανικά. Καλά, θα προσπαθήσω να το πω στα Αγγλικά. Εντάξει, αλλά να είστε λακωνικός παρόλα αυτά. Είπα λοιπόν ότι η πρώτη η πρώτη διάσπαση της συμφωνίας στο Κωσυφοπαίδιο προκάλεσε την Αυχαζία και την Οσετία. Μετά είχαμε την υπέρβαση της εντολής ε, του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, παρόλο που και εγώ ήμουν υπέρ της ανατροπής του Καντάφη. Αυτά ήταν τα δύο μηνύματα, τα δύο ξεκάθαρα χειρά μηνύματα που στείλαμε στη Ρωσία. Το τρίτο μήνυμα είναι η ε, δέσμευση να μην ε, επεκτείνουμε τις κάποιες δυνατότητες στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όταν έχουμε σχεδόν μια πολεοδομική επιχείρηση με επιμελητίες ε, ανάπτυξης, οποιοδήποτε ε, στρατιωτικός, ακόμη και χαμηλόβαθμος, γνωρίζει ότι το βασικό στον πόλεμο είναι η επιμελητιακή οργάνωση και όχι η οργάνωση επιτόπου. Γι' αυτό οδηγηθήκαμε στην κλιμάτωση. Συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την εδαφική ακαιρεότητα και ότι το ΝΑΤΟ είναι ακρογωνιαίος λίθος ε, για την άμυνα και την ασφάλεια. Αλλά το να δημιουργούμε ε, μια κατάσταση κρίσης και αντιπαράθεσης στην οποία προκαλούμε τις αντιδράσεις της Ρωσίας ε, χωρίς μια στρατηγική οργάνωση θα έχουμε όχι μόνο το τέλος της εταιρικής σχέσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας που ανήγγειλε ο κύριος Ράσμουσης, κάτι που είναι εξαιρετικά σοβαρό, αλλά θα έχουμε τη δημιουργία ενός άξονα κινέζικου και ρωσικού που θα έχει τεράστιες στρατηγικές σημασίες. Και δεν πάμε από ε, ε, μήπως ε, συσσωρεύοντας τις ε, νίκες της τακτικής θα διηγηθούμε σε μια στρατηγική ήττα σε τελική ανάλυση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρεκ Γιούρεκ, εκ μέρους των μεταρρυθμιστών συντονιστών, συγγνώμη για την υπέρβαση. Όχι, σέβομαι τον ιστορικό ρόλο της ΣΑΛΤΑ, αλλά τώρα εμείς είμαστε η τρίτη σε μέγεθος ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές μπορεί να αλλάξει η κατάσταση αργότερα. Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε η τρίτη σε μέγεθος ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση που προτιμώ να επανέλθω στην μητρική μου γλώσσα, την πολωνική. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι στην τελευταία ομιλία ο πρόεδρος Πούτιν δεν μίλησε για κυρώσεις, ούτε για αντίθετες κυρώσεις. Ε, ή μίλησε με πολύ ξεκαθαρούς πολιτικούς ρόλους. Μίλησε για αντιδράσεις και ανταπαντήσεις. Και αν θέλουμε να μας λάβει υπόψη σοβαρά και να πειράσουμε την ρωσική πολιτική, και εμείς δεν θα πρέπει να μιλούμε ε, σε επίπεδο κυρώσεων, αλλά να ε, βρούμε τις κατάλληλες αντιδράσεις. Είπαμε σωστά ότι η Ρωσία του, του Πούτιν ε, παραβίασε τη συμφωνία της ε, Βουδαπέστης ε, πριν από 20 χρόνια, πριν από, που έγινε πριν από 20 χρόνια. Ουσιαστικά όχι δεν την παραβίασε, αλλά την ακύρωσε. Και ε, από τη στιγμή που παραβιάστηκαν τα συμφέροντα της, της Δύσης από τη, και παραβιάστηκε η συνθήκη της Βουδα, Βουδαπέστης, αυτό έγινε από τη Ρωσία. Και αν εμείς δεν αντιδράσουμε και δεν παραβιάσουμε και εμείς αντίστοιχα την συνθήκη, τότε δεν θα μας λάβει υπόψη σοβαρά. Και δεν θέλουμε απλώς συμβολικές, αλλά πραγματικές αντιδράσεις, να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των πιο απειλούμενων συμμάχων του ΝΑΤΟ. Αλλιώς δεν θα μας, λάβα, θα μας λάβουν υπόψη σοβαρά. Και μάλιστα είχαμε την τελευταία σύνοδο κορυφή ε, που ήταν η συνέχεια του, του Βουκουρεστίου. Στο Βουκουρέστι δεν μιλήσαμε καν για συμβολική παρουσία του ΝΑΤΟ στις βαλτικές χώρες. Αν θέλουμε όμω επαναλαμβάνω, να μα λάβει σοβαρά υπόψη ο Πούτιν και θέλουμε να επηρεάσουμε τη ρωσική πολιτική, η παρουσία μα, η στρατηγική παρουσία του ΝΑΤΟ στι χώρε αυτέ, τη Βαλτική, δεν θα πρέπει να είναι απλώ συμβολική, αλλά ουσιαστική. Και αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα το ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν αμυντικό σύμμαχο. Θα πρέπει όμω να είμαστε σε θέση να προασπίσουμε του συμμάχου. Επίση, για την Εστονία είχε γίνει μια, ένα είδου επίθεση. Θα πρέπει να αντιδράσουμε με ένα γιατί δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη Ρωσία να επαναλάβει κάτι τέτοιο. Ποιο θυμάται σήμερα την Απχαζία παρόλο που δεν έχουμε αναγνωρίσει την απόσχησή της ε, από τη Γεωργία. Επίσης, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την ε, ταυτόχρονη παρουσία σας, δηλαδή και τον εκπρόσωπο της ΕΙΕΔ και του εκπροσώπου του ΝΑΤΟ. Γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε στενή συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και είναι εδώ θέμα αναγνώρισης της πραγματικότητας. Η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Είμαστε σύμμαχοι και δεν θα πρέπει να έχουμε επικάλυψη ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να μιλήσουμε για σωστό συντονισμό συντονισμό μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια και οι αναπτυξιακές δυνατότητες των χωρών μας. Ε, ε, δεν προτάθηκε από το ΝΑΤΟ αποκλεισμό της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να προτείνουμε τέτοιο αποκλεισμό. Γιατί αν δεν εγγυηθούμε καλύτερη παρουσία του ΝΑΤΟ στις Βαλτικέ χώρες, τουλάχιστον θα πρέπει να ζητήσουμε να αποκλειστεί η Ρωσία από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Επίσης θα πρέπει να έχουμε κοινή δράση σε διεθνεί οργανισμού και να μην ακολουθήσουμε δύο παράλληλες πολιτικές. Φυσικά σέβομαι ιδιαίτερος και τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, και ευρωπαϊκές χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Ιρλανδία ή η Αυστρία για παράδειγμα, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είναι απαραίτητος ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και των δύο οργανισμών. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λούζινγκ από την ΚΟΕ τώρα. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ σε κάποια σχόλια του προλαλήσαντος ο κύριος Πάσκου είπε κάθε βήμα, δυστυχώς έχει φύγει τώρα, κάθε βήμα που κάνουμε, κάθε κίνηση που κάνουμε θα πρέπει να είναι αντικειμενική. Δεν χωράει καμιά αμφιβολία. και οι συνάδελφοί μου στην πολιτική μου ομάδα έχουμε και εμείς πολύ κριτική στην πολιτική του Πούτιν να ασκήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική δράση ε, της Ρωσίας αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, και αναφέρομαι στην αποδοχή του κυρίου Γκάλερ. Είναι πολύ ασαφή τα πράγματα ακόμα και ξέρουμε σε ποιον όλουθρο μπορεί να μας οδηγήσουν και μας οδήγησαν στο Ιράκ εσφαλμένες παραδοχές που όλα αυτά που ακούμε ε, τα αμφισβητούν ε, απόστρατοι ή πρώην μέλη των μυστικών υπηρεσιών σε ανοιχτές επιστολές. Αυτό λέει γιατί τα αγνοούμε και τα ε, περιφρονούμε και δεν τα λαμβάνουμε υπόψη στη σκέψη μας. Και έχω συγκεκριμένη ερώτηση και παρατήρηση. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θέλω να φερθώ στις μονάδες ε, ταχείας επέμβασης. Κύριε η συνέχεια μιλάτε για εμπιστοσύνη. Εντάξει. Ε, ξεκινάμε από την παραδοχή ότι έχει καταχρηστεί την εμπιστοσύνη μας η Ρωσία και έχει διαταραχθεί αυτή η σχέση. Αλλά αυτές οι μονάδες ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ για μένα και αιχμή του δόρατος ε, είναι κάτι που μαθαίνω ότι θα χρησιμοποιείται παντού και στην Ανατολική Ευρώπη και όχι μόνο στο έδαφος της Συμμαχίας, αλλά αν έχουμε κρίσεις τύπου Ουκρανίας, που δεν είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, ε, μπορούν να δρουν, λέει, στα σύνορα με τη Ρωσία. Σωστά το ερμηνεύω έτσι. Και θέλω να ρωτήσω. Αυτό δεν είναι διάρρηξη της εμπιστοσύνης από δικής μας πλευράς, διότι υπάρχει υπόσχεση ότι δεν θα διευρυνθεί προς Ανατολά στο ΝΑΤΟ. Είναι μια υπόσχεση που έχει δοθεί στη Ρωσία στο παρελθόν. Και ρωτώ, κύριε Γκάλα, εγώ δεν σας διακόπτω ποτέ. Δημοκρατική λειτουργία έχουμε εδώ και θα σας παρακαλούσα να με αφήσετε να τελειώσω. Έλεγα λοιπόν ότι έχει ενδιαφέρον σε μια συζήτηση να βλέπουμε ποιος διακόπτει ποιον και ποια στιγμή. Δεν θέλετε να ακουστούν αυτά που λέω. Εάν θέλετε αφήστε με να μιλήσω με την ησυχία μου. Και ε, με τρόπο νυφάλαιο και αντικειμενικό να απαντηθούν αυτά παρακαλώ. Λοιπόν, ερωτώ. Συγγνώμη που μακρηγορώ, με διακόπτουν οι συνάδελφοι. Ε, δεν είναι επικίνδυνη αυτή η γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Δεν θεωρούμε πια ως εταίρο τη Ρωσία. Και λέμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία θεωρείται πλέον αντίπαλος του ΝΑΤΟ και όχι εταίρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσουβάρης από τους ε, πράσινους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Οι πράσινοι θέλουν να αποφύγουμε μια περαιτέρω στρατικοποίηση της ε, κρίσης στην Ουκρανία. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να γίνει από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Είναι μια πολύ ανησυχητική ε, εξέλιξη. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι θα πρέπει οι, <clears throat> οι κυρώσεις να θίξουν την ε, ρωσική οικονομία η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από τις εξαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου προς την Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει μια τέτοια λειτουργία των κυρώσεων. Επίσης η αποστολή της ΟΑΣΕ θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα εγώ λοιπόν να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην διαδικασία αυτή της πολιτικής αποστολής που έχετε αναφέρει. Κύριος Κωνσταντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά. Θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι τις αιτήσει που έγιναν από την κυρία Λόζιν για πρόσθετες πληροφορίες για τις πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να δοθούν σε σχέση με τις συγκεκριμένες κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας και επίσης θα ήθελα να έχω μια πιο συγκεκριμένη θέση από εσά για το κατά πόσο είναι βιώσιμη αυτή η επιλογή της Ουκρανίας και του Προέδρου Ποροσέγκο να αυξήσει τις αμυντικές και στρατιωτικές δαπάνες της τη στιγμή που υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η Ουκρανία αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να γνωρίζω ποιε μπορούν να είναι οι συνέπειε για τη χώρα αυτή αν σταματήσει η παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, τι θα σημαίνει αυτό για τον επόμενο χειμώνα στην Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ. Σαφχάουζεν από τους μη εγγεγραμμένους. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω καταρχήν κάτι το οποίο συνέβη την εποχή της ε, πτώσης του τείχους του Βερολίνου. Είχε υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των κεριών Κόλ και Μαζοβιέσκη να μην υπάρξει περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ Ξέρω ότι αυτό δεν είχε βέβαια επίσημο χαρακτήρα, ούτε κατεγράφει τις συμφωνίες τότε, αλλά υπήρχε μια σιωπήρη συμφωνία να μην διευρύνει το ΝΑΤΟ την παρουσία του στην Ανατολική Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω γιατί το ΝΑΤΟ και με ποιο δικαίωμα ασχολείται τώρα με τα θέματα της Ουκρανίας που η Ουκρανία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Επίσης θα ήθελα να πω στην κυρία Πρόεδρό μας ότι μέσα σε μία δίκη συνήθως υπάρχει διαδικασία κατά αντιμολία, να είναι παρόντες και οι δύο πλευρές. Θα ήθελα να έχουμε τη δυνατότητα να προσκαλέσουμε τον Ρώσο πρεσβευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρουσιάσει τη δική τους άποψη των πραγμάτων. Επίσης, θα ήθελα να υπάρχουν και κάποια ερωτήματα προς τον Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Μιλάει για χιλιάδες Ρώσων στρατιωτών. Μήπως είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό το οποίο αναφέρουμε για τη Λιβύη, ότι έχουμε Ρώσους τζιχαδιστές μέσα σε εισαγωγικά, είναι δηλαδή απόστρατοι παλιοί στρατιώτες οι οποίοι εθελοντικά κατά κάποιο τρόπο μέσα σε εισαγωγικά και πάλι συμμετέχουν στη σύραξη αυτή όπως οι εθελοντές μέσα σε εισαγωγικά που παρέχει η Τουρκία στην ε, Συρία θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν αν είναι πραγματικά στρατεύματα ή αν είναι ε, κάποιο είδος εθελοντών κατά κάποιο τρόπο. Αν ήθελε πραγματικά η Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία θα το έκανε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Χιλιάδες ατόμων λοιπόν δεν είναι χιλιάδες στρατιώτες. Δεύτερον σε ό,τι αφορά την εδαφική ακαιρεότητα. Εσείς γνωρίζετε ότι έλαβε χώρα ένα πραξικόπημα στην Ουκρανία και όταν μιλάμε για εδαφική κυριαρχικότητα υπήρξε μια ουσιαστική ρήξη σε σχέση με τις συμφωνίες που είχαν υπογραφεί με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναγκάστηκε να παρετηθεί. Ουσιαστικά έχασε την εξουσία του. Εδώ βρίσκεται μια ιδιαίτερη κατάσταση που δεν έχει να κάνει με, το, με τη φυσιολογική κατάσταση του διεθνούς δικαίου. Έχουμε μια ρήξη σε σχέση με την ιστορική συνέχεια του Ουκρανικού κράτους. Και θέλω να θέσω το ερώτημα γιατί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ Κωσόβου και Βοσνίας Ερζεγοβίνης και της Ουκρανίας. Γιατί δεν μπορεί και το ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας να αποκτήσει μια εδαφική κυριαρχικότητα. Τρίτον, θέλω να θέσω το εξής ερώτημα σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό των κρατών μελών και της Ρωσίας Γνωρίζετε το Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ότι ο στρατιωτικός προϋπολογισμός των κρατών μελών ξεπερνάει τον προϋπολογισμό και της Ρωσίας στο στρατιωτικό και τον ίδιο τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν τα πράγματα στα σωστά τους μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Only one intervention. Παρακαλώ, οι επόμενε ομιλίε θα είναι ενός λεπτού μόνο. Ο κύριο Έλερ, τα μέλη του Προεδρείου έχουν τώρα τη σειρά. Παρακαλώ, ένα λεπτό κύριε Έλερ. Um, Μια σύντομη ερώτηση μίλησαν οι πολιτικέ ομάδες οι συντονιστέ. Τι θέλετε. Ε, άλλοι μιλούν πέντε λεπτά και άλλοι μιλούν ένα όμω. Κύριε Έλερ, το λόγο. Μια σύντομη ερώτηση έχω. Μιλήσατε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και στον κυβέρνο χώρο στην Ουκρανία ε, είναι μια κατάσταση ασύμετρου πολέμου με χερσαία στρατεύματα ρωσικά που δεν είναι επισήμως ρωσικά και όλο και περισσότερες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Δεν θα το χαρακτήριζα πόλεμο, αλλά είναι υψηλή εντάσεως δράση στο διαδίκτυο. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς απαντήσουν είναι σχετικά περιορισμένη η απόκρισή μας. Το σκεφτόμαστε αυτό, γιατί Αναφερθήκατε ιδιαίτερα στην ασφάλεια στο διαδίκτυο. Πώς θα μπορούσατε να την εξασφαλίσετε, γιατί υφίστανται επιθέσεις από την FSB και ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ κύριο Στετίνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δοθεί απάντηση στην ερώτηση που υπέβαλα προηγουμένως. Ο κύριος Λαντσμπέργης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να έρθει εδώ ο Ρώσος πρέσβης. Ε, ακούσαμε τη ρωσική θέση πολύ ωραία από κάποιους συναδέλφους να περιγράφεται. Δεν χρειάζεται να καλέσουμε τον πρέσβη. Ε, να σας ενημερώσω για κάποιες νέες εξελίξεις. Few, few new λέω κάποιες νέες εξελίξεις ε, που έγιναν στη Βαλτική πρόσφατα. Πρώτον, ένας ε, ε, στον όσο αξιωματικός συνελήφθη απήχθη σε στονικό έδαφος και αν κατάλαβα καλά ήταν επιχείρηση του Κρεμλίνου που έγινε σε επικράτεια ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγωγή αξιωματούχου, δεν ήταν αξιωματικός, ήταν ε, πολίτης ε, και δεν ήταν σε επιχείρηση σε εχθρικό ή αλλοδαπό έδαφος. Συζήτησα με κάποιους εστωνούς συναδέλφους ε, και η αντίδρασή τους ήταν κάπως χλιαρή για να μην πω τίποτα χειρότερο. Και είπαν ότι είναι κατάσκοπος, τη δουλειά του κάνει και τι να κάνουμε, αυτό είναι το τμήμα της δουλειάς. Και τι εμείς θα κάτσουμε έτσι με σταυρωμένα τα χέρια και να μας απαγάγουν τους ανθρώπους μας και να τους ε, πηγαίνουν στη Μόσχα. Επίσης, η Ρωσία απείλησε να προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά των Λιθουανών που ανήθηκαν πριν από 25 χρόνια να καταταγούν στο Σοβιετικό στρατό, στο Ρωσικό τότε. Το ξέρω ότι είναι μεγάλα λόγια αυτά, αλλά ουσιαστικά σημαίνει απαγόρευση θεώρησης διαβατηρίων για κάποιες χιλιάδες Λιθουανούς, συμπατριώτες μου. Ερωτώ λοιπόν, ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά. Βεβαίως μιλάμε για αποκλιμάκωση και τα λοιπά, αλλά εγώ πιστεύω γενικά ότι τώρα πρόκειται για κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Οπότε, ποιο είναι το μήνυμα που θα πρέπει εμείς να εκπέμψουμε στις χώρες μας από τις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παρνιό. Ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα μια φράση να πω και ήταν απόδειξη ότι φαίνεται ότι η γαλλική ακραδεξιά έχει γίνει ε, πρόσωπος του κυρίου Πούτιν. Ε, είπαμε ότι θα πρέπει να ε, δραστηριοποιηθούμε για να εξασφαλίσουμε την εδαφική αικαιρεότητα της Ουκρανίας. Ναι, είπαμε ότι θέλουμε διαφορετική εντολή σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Ναι, και έχουμε δίκιο πιστεύω κύριε Πρέσβη. Είπαμε να εφαρμόσουμε τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ουκρανία και να αναγγείλουμε και την προετοιμασία της, έκθεση, της έκθεσης μας για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και επίσης να ενισχύσουμε τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας προκειμένου να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ ε, της στρατιωτικής πλευράς που εκπροσωπείται από τον ΝΑΤΟ και της διπλωματίας και της πολιτικής δράσης ε, που εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΥΠΑ της εκπροσώπου αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αρχική κρατών και κυβερνήσεων να συνειδητοποιήσουν ότι η δημοσιονομική δέσμευση υπέρ μιας ε, ε, αποτελεσματικής άμυνας ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί δεν θα πρέπει να βρισκόμαστε πάντα υπό την αιγύδα του ΝΑΤΟ να μπορούμε και εμείς μόνοι μας να επιταχύνουμε τις διαδικασίες γιατί και εμείς ως ευρωβουλευτές και μέλη της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνα, θα πρέπει να αρχίζουμε να σφυριλατούμε τη δική μας στρατιωτική επιχείρηση φυσικά στα πλαίσια των ε, ευρωπαϊκών οργανώσεων και φορέων. Η κυρία Γκόμε, ευχαριστώ. Και εγώ ε, θα προτιμούσα να ακολουθήσουμε απευθείας του Ρώσο πρέσβη παρά να ακούμε τους εκπρόσωπους της ακροδεξιάς του Λεπέν στη θέση των μισθοφόρων του Πούτιν. Ο κύριος Γερασίμοφ το Φεβρουάριο του 2013 δημοσίευσε κάτι αναγγελίες γιατί πού είναι το πρόβλημα, δεν λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τη Ρωσία ή έχουμε πρόβλημα μυστικών υπηρεσιών. Και τι γίνεται με τις τρέχουσες πρόκλησεις ε, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κυρώσεων από πλευράς της Γαλλίας ή να προετοιμαστούμε για την επόμενη ρωσική κίνηση. Κύριε Πατουράη, μιλήσατε σωστά για τις ε, πολλές επιπτώσεις ε, της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Αναφερθήκατε και στην Κρυμαία, που είπατε ότι αυτό δεν σήμαινε αλλαγή απλώς των σύνορων, αλλά ε, για παραβίαση της ε, ε, συνθήκης της για τα πυρηνικά και την εξασφάλιση της προστασίας από τους πέντε μετά τον πυρηνικό αφοπλισμό της Ουκρανίας. Και υπήρξε και το θέμα της αποτροπής ε, χωρών όπως το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και άλλων χωρών που δεν έχουν προσυπογράψει συμφωνία για τα πυρηνικά, Πακιστάν και Ισραήλ. Τι σημαίνει όμως, ε, τι σημαίνουν οι δηλώσεις της Ρωσίας ότι θα, ε, θα επενδύσει στα πυρηνικά και στην πυρηνική ενέργεια και ποια θα είναι η αντίδραση των μελών του ΝΑΤΟ. Θα ξεκινήσει μια νέα κούρσα των πυρηνικών εξοπλισμών. Ξέρουμε ότι τα πυρηνικά δεν έχουν καν αποτρεπτικό ρόλο. Ή μήπω έτσι θα στερηθούμε πόρους που χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως ε, πολύ πιο δραστικά για να ε, ενισχύσουμε την άμυνά μας ε, κατά της πιθανής ρωσικής επίθεσης. Είπατε ότι τα συμπεράσματα του Κάρντιφ έδειξαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία για τον ΝΑΤΟ ποτέ και η δυνατότητά της στα πλαίσια ασφάλειας και άμυνας το ίδιο. Όμως ε, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο ύψος των περιστάσεων και από πολιτική και από πρακτική άποψη. Τι νόημα έχει ο κύριος Μπαρόζο να υποκύπτει στις απειλές του κυρίου Πούτιν και μάλιστα ε, αποκαλύφθηκαν οι πληροφορίες που έλεγε ότι σε δύο εβδομάδες θα είναι στο Κιεφ. Γιατί έπρεπε να φοβάται ο κύριος Βαρόζο να αποκαλύψει αυτές τις ε, συνομιλίες. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα μιας τέτοιας κατάστασης. Ο κύριος Κούζο. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι. Παρακαλώ να είστε σύντομος, λέει η πρόεδρο. Καταρχήν θέλω να επαναλάβω αυτό που έλεγε η Σαμπίνε. έχουμε ένα πολεμικό λόγο που ακολουθείται από τους περισσότερους ομιλητές. Αλλά εμείς θεωρούμε τα τελευταία 25 χρόνια το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνει το ΝΑΤΟ είναι να αυξήσει τις στρατιωτικές της ικανότητες. Η δική μου χώρα συμμετέχει εκεί. Τονίστηκε τότε ότι παραγωγικά υπήρχαν οι πύραυλοι του Ιράν που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε μια στρατιωτική απάντηση από το ΝΑΤΟ, ενώ οι μυστικές υπηρεσίες λέγανε ότι δεν έχουν εμβέλεια πάνω από 2.000 χιλιόμετρα και τότε είχαμε στρατιωτική συνεργασία με τη Ρωσία. Επίσης το θέμα της διεύνησης του ΝΑΤΟ, το οποίο ουσιαστικά παραβιάζει την ε, συμφωνία για τις σημαντικές δυνάμεις στην ε, Ευρώπη. Κύριε Πατουράη, φταίει η Ρωσία ή ουσιαστικά έχει ενώπιον της ένα νέο αντίπαλο που είναι το ΝΑΤΟ όπως έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Μήπως θεωρείτε ότι η αύξηση των ε, δυνάμεων ταχείας αντίδρασης ή οι βάσεις γύρω από τη Ρωσία δεν προωθούν τα πράγματα σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Μήπως θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κλιμάκωση των πραγμάτων. Η Ρωσία είναι στην Ευρώπη. Είναι γείτονά μας. Γιατί να έχουμε αυτή την ένταση. Γιατί εμείς να πιέσουμε τη Ρωσία προ αυτή την κατεύθυνση. μήπω ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα συγχαίρονται με τα αμερικανικά σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ κύριο Συναδεινό και μετά ο πρέσβης ε, που πρέπει να φύγει. Ευχαριστώ. Θα, δεν θα αναφερθώ στην ε, Ρώσο-Ουκρανική κρίση κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, αλλά για κάποιο θέμα το οποίο άρτεται της ε, πατρίδος μου Ελλάδος. Στην ε, σύνοδο κορυφής λοιπόν προσφωνήθηκε ο Υπουργός της ΦΥΡΟΜ ως Υπουργός της Μακεδονίας. Πιστεύω ότι αυτό έγινε εκ παραδρομής και όχι εσένα. Sorry, sir. Συγγνώμη κύριε, είμαι υποχρεωμένη να σας διακόψω. Έχουμε θέμα στην ημερήσια διάταξη και μιλούμε για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Έχουμε άλλο θέμα αμέσως μετά που θα συζητήσουμε τη σύνοδο κορυφή του ΝΑΤΟ και εκεί θα μιλήσετε. Το λόγο έχει ο κύριος Ποπόφσκι. Uh, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ορισμένα από τα ερωτήματα απευθύνθηκα στο James, θα απαντήσω εγώ στο δικό μου σκέλος και από δική μου πλευράς. Για το στόχο των ε, αμυντικών δαπανών δεν έχουμε αριθμητικό στόχο, αλλά ο στόχος αυτός καθ' αυτός έχει σημασία μεν, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η διάρθρωση και η δομή του 2% που διοχετεύεται αυτό. Στο ΝΑΤΟ το 20% ζήτησαν για τον εξοπλισμό. Ξέρουμε ότι περισσότερες χώρες, τα κράτη-μέλη της Ένωσης, ε, δαπανούν το 60% των ε, αμυντικών δαπανών στο προσωπικό και όχι στην ενίσχυση των ικανοτήτων. Βεβαίως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας για να διευκολύνουμε κάπως ε, μια, ένα ελαφρύ συντονισμό για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού για να φτάσουμε κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. γίνει μια ερώτηση για το αν απέτυχαν οι μυστικές υπηρεσίες. Ε, δεν είναι δικός μου ρόλος να απαντήσω. Δεν έχουμε εμεί δυνατότητες και ικανότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, μυστικών υπηρεσιών, εκτός από το κέντρο αυτών ε, πληροφοριών, που είναι ένα κέντρο που συγκεντρώνονται εκεί πληροφορίες που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αλλάξει η αντίληψη για την απειλή στην Ευρώπη. Ήδη πριν από ένα χρόνο, ή και δύο χρόνια, Πολλά από τα ανατολικό ευρωπαϊκά κράτη ε, είχαν κατηγορηθεί ότι ήταν υπερβολικοί στους φόβους τους για τη Ρωσία. Ε, αυτό πια δεν ισχύει. Έχει αλλάξει πια η αίσθηση για την απειλή. Μπορεί να γίνεται με βραδείς ρυθμούς, αλλά αλλάζει. Γιατί υπάρχουν τα στοιχεία εδώ. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ε, αντικατοπτρίζεται και στη νέα εκτίμηση και αξιολόγηση της ύπατης εκπροσώπου που θα κατατεθεί. Τώρα, για τις κυρώσεις και την κλιμάκωση. Είναι δύσκολο να τραβήξει καμία γραμμή, να πει που θα σταματήσουμε. Έχουμε κάνει πρόοδο για κάποια πρόσωπα που κατηγορήθηκαν ε, ότι παραβιάζουν την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Ήταν η δεύτερη φάση και τώρα είναι η τρίτη φάση με οικονομικές κυρώσεις ε, ε, σοβαρές που δείχνουν αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα καμιά φορά φαίνονται αργότερα, αλλά τώρα υπάρχουν ροές κεφαλαίων από τη Ρωσία, διαφυγή κεφαλαίων μέχρι 100 δις ευρώ ε, πιέζεται το ρούβλι, μειώνεται ο τουρισμός ε, των Ρώσων και υπάρχουν και άλλα στοιχεία ότι ε, αποδίδουν οι κυρώσεις αλλά έχουν και ένα αντίτιμο με αντίπεινα της Ρωσίας που πλήττουν πολύ τα δικά μας κρατη και χρειάζεται αποζημίωση εκείνων που έχουν υποστεί ζημίες γιατί έχουν χάσει την πρόσβασή τους στη ρωσική αγορά ο πόλεμος στον κυβερνοχώρο στην Ουκρανία. Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων μονάδων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του πολέμου στο διαδίκτυο, αλλά μπορούμε να ενισχύσουμε την αντίσταση ε, μέσω δημιουργίας ε, θεσμών και υποδομών γενικότερα. Ε, όταν κάνουμε μια συνεργασία πολιτικών δομών με στρατιωτικές ή απλώς υποστήριξη δημιουργίας κρατικών θεσμών, ε, μπορούμε να ασχοληθούμε και με αυτές τις επιθέσεις στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή της στις εμμενικές δαπάνες ε, δεν μπορούμε παρά να βελτιώσουμε εκεί την απόδοσή μας μέχρι τον Ιούνιο του 2015 ε, και το επόμενο Συμβούλιο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων που θα συζητήσουν αυτά τα θέματα με τη νέα ε, ε, ομάδα στην υπηρεσία εξωτερική δράση θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά σε ό,τι αφορά τι στρατιωτικέ δαπάνε αυτές καθ' αυτέ και τη μεγαλύτερη συνεργασία για να στηθεί αυτό χρειάζεται περισσότερο χρόνο και δεν θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ βραχυπρόθεσμα ε, αποτελέσματα, τουλάχιστον όχι μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία. Η νόμιμα εκλεγμένη Ουκρανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος μάλλον ε, υπέγραψε αυτή τη συμφωνία. Δεν υπάρχουν νομικά προσκόμματα, είναι σαφέστατη η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Ε, κύριε Πατουράη, παρακαλώ, ε, Ευχαριστώ. Θα είμαι όσο πιο συνοπτικός γίνεται. Έμαθα τρία πράγματα. Καταρχήν ότι ε, οι συνεδριάσει εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσε από ό,τι στο ΝΑΤΟ. Θα προσπαθώ να έρθω όσο πιο συχνά γίνεται. Δεύτερον, το πιο δύσκολο έργο στον κόσμο είναι να κρατά, επιβάλλει την πειθαρχία στους ευρωβουλευτές. Δεν φανταζόμουν ότι ήταν τόσο περίπλοκο αυτό το έργο. Και επίσης ε, συμφωνώ με την ε, θετικό απολογισμό που έκανε ο κ. Σποπόφσκι. Ε, και ότι ίσως ο λόγος που εμφανίζεται τόσο συχνά στο τελευταίο ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γιατί πρώτη φορά έχουμε τόσο μακροσκελές ανακοινωθέν. Αλλά αυτό πραγματικά δείχνει και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών. Κάτι που ακούσαμε από πολλούς είναι γιατί δεν, ε, είχαμε, γιατί δεν λάβαμε υπόψη την περίφημη ε, ομιλία του κυρίου Γερασίμοφ, ε, του αρχηγού του ΓΕΘΑ, Φαντάζομαι πολύ έχετε σπουδάσει διπλωματία και είχα μάθει κι εγώ ότι για να καταλάβει κανείς τη Ρωσία θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι είναι ένα ένιγμα τυλιγμένο μέσα σε ένα πάζλ. Η πείρα μου όμως με έχει δάξει το αντίθετο, ότι ε, λένε ακριβώς τι θα κάνουν και κάνουν ακριβώς αυτό που λένε. Απλώς εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε και ε, αυτό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα, ότι φαίνεται ότι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι η Ρωσία θα κάνει αυτό που λέει. Και μετά το κάνει και μετά ε, εκπληθόμαστε και δεν θέλουμε να πιστέψουμε για το επόμενο τους βήμα. Και αυτό έχουν δείξει τα νομοθετήματα που έχουν περάσει από το, από το Ρωσική Βουλή που δίνει τη Μόσχα στο δικαίωμα να επεμβαίνει ακόμη και στρατιωτικά όταν α, θεωρεί ότι απειλούνται τα συμφέροντα της ακόμη και για ιστορικά εδάφη της Ρωσίας. Κάτι που οδηγεί σε ανατροπή των συνόρων και το δικαίωμα στα σύνορά σας. Αν έχετε ιστορικά ε, και ο τρόπος που δίνει τα διαβατήρια σε μειονότητες σε άλλες χώρες ε, όπως το κάνει είναι χαρακτηριστικά. Όλα αυτά είναι πολύ αποσταθεροποιητικά. Και συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να διαβάζουμε αυτά που λένε οι Ρώσοι, να διαβάζουμε τις νομοθεσίες τους, ε, να τα πιστεύουμε και να προετοιμαζόμαστε ανάλογα. Και επίσης αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε αντιπαράθεση ή κλιμάκωση. Κάτι τέτοιο το απευχόμαστε. Και θα ήθελα να απαντήσω στην ανησυχία που εξέφρασα με μερικοί ότι έχουμε κλιμάκωση, αν κοιτάξουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ δεν είμαι βέβαια ούτε από Ευρωπαϊκή χώρα, ούτε είμαι Ευρωπαίος, ε, προσπάθησαν σκληρά οι χώρες ε, να φέρουν τη Ρωσία στο σύστημα και στις δομές. Όχι μόνο στην ευρωατλαντική ασφάλεια και συνεργασία ευρωπαϊκή, αλλά και στην παγκόσμια συνεργασία. Και σεβόμαστε το βάρος και τη σημασία της Ρωσίας και δημιουργήσαμε και Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Είναι η μόνη χώρα που έχει ίση ψήφο με τους συμμάχους, η Ρωσία. Δεν έχουμε δώσει τέτοιο δικαίωμα σε καμία άλλη χώρα εταίρο με ένα πλέγμα υποεπιτροπών, στις οποίες επίσης έχει δικαίωμα ίσης ψήφου η Ρωσία. Έχουμε το G7, το G20, την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου και ούτω καθεξής. Ολόκληρος ο κόσμος προσπάθησε να εντάξει την Ρωσία στο σύστημα και να προσαρμόσει το σύστημα ώστε να σέβεται τη Ρωσία. Αυτό που βλέπουμε όμως σήμερα είναι ότι μία τέτοια τακτική δεν απέφερε καρπούς και αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε συζητήσει με τη Ρωσία και σχέση με τη Ρωσία, ώστε να αισθάνεται, αυτό το σεβασμό η Ρωσία, αλλά να ε, γίνονται σεβασμό, σεβαστές και οι δικές μας ε, αρχές ε, νομοθεσίες και το δικό μας σύστημα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ειρήνη, η σταθερότητα και τα σύνορα στην Ευρώπη είναι οι βασικές αρχές, δομές και διαδικασίες που πρέπει να προσπίσουμε. Και αν τα ρωσικά συμφέροντα αντιβαίνουν σε αυτού τους νόμους, τότε έχουμε πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα το δημιουργεί η Ρωσία και όχι εμείς. Και δεν θα πρέπει εμείς να υπομοιζόμαστε την ευθύνη ε, όταν παραβιάζονται αυτά τα όρια. Γιατί είναι συγκεκριμένες οι νομοθεσίες, οι νομοθετικέ διατάξει που θα πρέπει να τηρηθούν. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε καλύτερη ασφάλεια στα μέλη μας, ε, στα κράτη-μέλη, όσο συνεχίζεται η κλιμάκωση. Και είναι αναφυσβήτητο ότι το ΝΑΤΟ δύναται και οφείλει να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ε, μελών της. Αυτό όμως με μέτρο και όχι με τρόπο που θα προκαλεί την κλιμάκωση. Και όπως αναφέρθηκε, δεν αναπτύσσουμε ε, σημαντικό αριθμό μονίμων στρατευμάτων στις βαλτικές χώρες στην Πολωνία. Έχουμε μόνο μικρές δυνατότητες ε, υποδοχής ε, μη μάχημες, ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε στη συνέχεια στρατιωτικές δυνάμεις, αν κάτι τέτοιο αποβεί απαραίτητο. Και κάτι τέτοιο είναι πολύ λογικό και εντάσσεται πλήρως ε, στις δεσμεύσεις που έχει κάνει το ΝΑΤΟ και στους υπόλοιπους. Και δεν είναι θέμα όποια σχέση και αν έχει μια χώρα μέλος με τη Ρωσία, κανείς δεν πιστεύει ότι παραβιάζονται οι δεσμεύσει που έχει κάνει το ΝΑΤΟ απέναντι στους συμμάχους του. Επίσης, τέθηκε το θέμα των βαλτικών χωρών. Προσωπικά δεν έχω καμία αφιβολία ότι αν οι βαλτικέ χώρε και τα νέα μέλη του ΝΑΤΟ δεν, ήταν, δεν είχαν προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ, θα αντιμετώπιζαν πολύ μεγαλύτερε δυσκολίε. Βρίσκονται σε ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον και θα είχαν μεγάλε δυσκολίε να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Και είναι σημαντικό να εγγυηθούμε την ασφάλεια αυτών των νέων μελών. Είναι θέμα ευρωπαϊκής ασφάλειας και όχι μόνο δικής τους ασφάλειας. Και αυτό ισχύει όχι επειδή είναι μέλη μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επειδή είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και θα πρέπει να χαιρετήσουμε αυτό το γεγονό και να μην, μα απασχολεί. Τώρα, θα πρέπει να διαψεύσουμε του μύθου ε, για δεσμεύσει που έχει αναλάβει το ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Όχι. Δεν υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσει. Μπορεί να έγινε κάποιε παρασκηνιακέ συνομιλίε, ε, αλλά δεν τι γνωρίζω. Ουδέποτε ε, είτε το ΝΑΤΟ είτε κάποιο κράτο δεν έχει αναλάβει δεσμεύσει, Γιατί το άρθρο 10 του καταστατικού χάρτη προβλέπει ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ε, δημοκρατία που πληρεί τι προδιαγραφέ του ΝΑΤΟ έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη. Δεν έχουμε αναλάβει δέσμευση για μη διεύρυνση ουδέποτε. Οπότε αυτό είναι ένα επιχείρημα του Κρεμλίνου και θα πρέπει να σταματούμε να το χρησιμοποιούμε εμεί οι ίδιοι, γιατί δεν ευσταθεί, ουδέποτε δεν αναδόθηκαν τέτοιε δεσμεύσει. Τώρα, για πραγματικά στοιχεία σε σχέση με την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων. Έχουμε στοιχεία για ανάπτυξη τακτικών στρατιωτικών τμήματων στην Ουκρανία και έχουμε δημοσίευσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της πληροφορίας, οπότε μπορείτε να τα δείτε. Μιλάμε για μερικές χιλιάδες, τρεις χιλιάδες, ίσως λίγο παραπάνω. Τώρα έχει μειωθεί αυτός ο αριθμός. Υπήρξαν και ειδικέ δυνάμεις των ε, Ρώσων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Υπήρξε στρατιωτικός εξοπλισμός ο οποίος ε, εισήλθε στην Ουκρανία, υπήρξαν ε, ιδιωτικές ε, δυνάμεις ασφαλείας που χρησιμοποιούν πρώην στρατιωτικούς που ήταν όπως είπανε σε διακοπές μέσα σε εισαγωγικά. Αυτή ήταν μια από τις εξηγήσεις που μας δόθηκαν. Όταν λέτε να είμαστε σοβαροί, ναι, είμαστε σοβαροί. Πράγματι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε καλύτερη σχέση με τη Ρωσία. Θέλουμε και το τονίσαμε. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση η οποία επικρατεί, είτε μα αρέσει είτε όχι. Προσπαθούμε εδώ και 20 χρόνια να φτιάξουμε καλύτερη εταιρική σχέση με τη Ρωσία, αλλά τώρα είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση την οποία την προκαλέσαμε εμεί. Για τις κυρώσεις αυτό είναι ευρωπαϊκό θέμα, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί τώρα να επιβάλλει σε κανένα κυρώσεις. Η κατάσταση της Εστονίας είναι πολύ δύσκολη. Καταλαβαίνω ότι η εστονική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα σε διμερή βάση. Αυτό είναι δική τους απόφαση. Τη σεβόμαστε. πυρηνική, κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών. Το ΝΑΤΟ έχει μειώσει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων που έχουμε στο προστάσιό μας στις χώρες του ΝΑΤΟ. Και στην Ευρώπη συγκεκριμένα κατά 90% έχει μειωθεί το πυρηνικό προστάσιο του ΝΑΤΟ. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως ξέρετε μαζί με τη Ρωσία προσπαθούν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τα, τις στρατηγικές πυρηνικές κεφαλές. Και δεν υπάρχουν πια τακτικά πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχει μια σαφής πολιτική του ΝΑΤΟ ότι τα πυρηνικά όπλα παραμένουν βασικό στοιχείο της δύναμης αποτροπής του ΝΑΤΟ. Δεν έχουμε λοιπόν σχέδια να αυξήσουμε τον αριθμό τους και υπήρξαν πολλές προσπάθειες να μειωθεί ο αριθμός των πυρηνικών όπλων και έχουν γίνει πραγματικά μειώσεις, αλλά η αποτροπή πυρηνική είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής του ΝΑΤΟ και σε αυτό περιλαμβάνονται και τα πυρηνικά όπλα. Και όπως είπατε, σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στα συμβατικά όπλα, αλλά τα πυρηνικά παραμένουν. Σας ευχαριστώ κύριε Αναπληρωτή Γενική Γραμματέα. Μπορώ να κλείσω λοιπόν αυτό το σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ τον ε, πρέσβη Ματσέη Ποπόσκι για την παρουσία του στην συνεδρίασή μας και για την ε, πλήρη παρουσίαση που μας έδωσε τόσο σε ό,τι αφορά τη συνάντηση των Υπουργών ε, Άμυνα, την Άμυνη Σύνοδο Υπουργών, την άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνα και για τα θέματα επίση Ουκρανία. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη. Ο κύριος ε, Απατουράη θα είναι ο κύριο Ομιλητή και θα μας πληροφορήσει για τα συμπεράσματα της ε, πρόσφατης συνόδου του ΝΑΤΟ στο Νιούπορτ. Έχετε το λόγο κύριε Πατουράζη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συζητήσαμε ένα από τα κύρια στοιχεία αυτής της Συνόδου που ήταν η κρίση της Ουκρανίας και όλα αυτά τα οποία σημαίνουν αυτές οι καταστάσεις για τον ΝΑΤΟ. Θα ήθελα εδώ να σταθώ σε κάποια από τα άλλα στοιχεία της Συνόδου Κορυφής που μπορεί να ενδιαφέρουν τους συναδέλφους σας. Ένα θέμα είναι το Αφγανιστάν συζητήθηκε αυτό διαμακρών. Είχαμε μια χωριστή συνάντηση για το Αφγανιστάν με τους εταίρους μας της ΙΣΑΦ. Όπως ξέρετε η αποστολή ΙΣΑΦ, η αποστολή αυτή της στρατιωτική του Αφγανιστάν φτάνει στο τέλος της. Είχαμε προετοιμασία για την περίοδο μετά από το 2014 τρεις γραμμές υποστήριξης για το Αφγανιστάν. Καταρχήν μια μικρότερη συμβουλευτική και εκπαιδευτική δύναμη, το Resolute Support όπως λέγεται, Δεύτερον, μια μεγάλη χρηματοδότηση, 46 δισεκατομμύρια ευρώ, για να υποστηρίξουμε τις στρατιωτικές δυνάμεις του Αφγανιστάν στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, γιατί είναι φανερό ότι δεν μπορούν αυτοί να υπομισθούν το κόστος της ε, αμυνάς τους. Είναι πολύ πιο φτηνό να έχουμε λοιπόν τις ε, δυνάμεις, για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ να υποστηρίζουν οικονομικά τις αφγανικές δυνάμεις παρά να στέλνουν δικούς τους στρατιώτες και επίσης θα πρέπει να έχουμε μια μετάβαση στη σχέση μας με το Αφγανιστάν ώστε το Αφγανιστάν από θέατρο στρατιωτικών επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει ένας πολιτικός εταίρος. Έχουμε πάνω από 40 τέτοιου είδους ε, συμφωνίες συνεργασίες με χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και έχουμε ένα φυσιολογικό πολιτικό διάλογο με τις χώρες αυτές. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και να έχουμε μια μετάβαση από την στρατιωτική σχέση. Η δυσκολία είναι τώρα βέβαια το εσωτερικό πολιτικό στερέωμα στο Αφγανιστάν που είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και επειδή δεν έχει επιτευχθεί ακόμα στο Αφγανιστάν η δημιουργία μιας κυβέρνησης δεν έχουν ακόμα υπογράψει τις απαραίτητες νομικού χαρακτήρα συμφωνίες για την παρουσία διεθνών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Εάν δεν το κάνουν τώρα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, τότε για λόγους τεχνικούς, όπως και στην περίπτωση του Ιράκ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό της αποχώρησης όλων των διεθνών δυνάμεων από το Αφγανιστάν. Δεν θέλω να παραλληλήσω ιδιαίτερα την κατάσταση του Αφγανιστάν με αυτή του Ιράκ, αλλά η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι αυτό δεν ήταν μια θετική εμπειρία. Πιστεύω ότι το Αφγανιστάν θα πρέπει να έχει συνεχή διεθνή υποστήριξη. Πιστεύουμε όσο πιο γρήγορα μπορεί να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση και γίνουν οι απαραίτητε νομικέ ρυθμίσει, τόσο το καλύτερο θα είναι και για το Αφγανιστάν και για μα. Αλλά φυσικά δεν εξαρτάται από εμά αυτό. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο στη Σύνοδο Κορυφή ήταν η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Ε, μια ορολογία που δεν θα πρέπει να αποδεχτούμε. Μπορεί αυτοί να λένε ότι είναι ένα κράτος αλλά δεν είναι κράτος. Ουσιαστικά τους δίνει μεγάλη, μεγαλύτερη ε, ακτινοβολία από ό,τι αξίζουν. Εν πάση περιπτώσει αυτή η ομάδα, αυτό το μόρφωμα είναι μια άμεση απειλή για όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό και οι ακρότες που έχουν κάνει στη Συρία και το Ιράκ είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών οι οποίοι πολεμούν σε αυτό το μόρφωμα είναι ξένοι για τις περιοχές αυτές και έρχονται από την Ευρώπη, όχι από το Βέλιο, συγκεκριμένα από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Και στη Σύνοδο Κορυφής της υπήρξε μεγάλη ανησυχία για την ανασφάλεια που μπορεί να προκύψει είτε υπομορφή μιας άμεσης ανθρωπιστικής κρίσης και δεύτερον η δυνατότητα να υπάρχει μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση της περιοχής αυτής και τρίτον ο κίνδυνος ότι αυτοί οι ξένοι ε, μαχητές μπορούν να αποτελέσουν μια απειλή και για τη Δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει μια συνένεση ότι αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα θα έχουμε πράγματι τρομοκρατικές επιθέσεις στις χώρες μας από αυτές τις χιλιάδες μαχητών του Ισλαμικού κράτους που έρχονται από την Ευρώπη και οι οποίοι μπορεί να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη κάνουν μεγάλες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Αυτό ήταν πάντως ένα θέμα που συζητήθηκε στην Ουαλία και είδατε τώρα σήμερα ο πρόεδρος Ομπάμα στην ομιλία του τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια συμμαχία για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και εδώ το ΝΑΤΟ μπορεί να παίξει ένα υποστηρικτικό ρόλο. Έχουμε μια συμφωνία εταιρική σχέση με το Ιράκ και είχαμε μια αποστολή εκπαίδευση εκεί στο Ιράκ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι αντίστοιχο για το Ιράκ και το ΝΑΤΟ μπορεί να παίξει ένα συντονιστικό ρόλο για διάφορες μορφές υποστήριξης που δίνουν οι σύμμαχοί μας σε διμερή, ε, διμερές επίπεδο για το Ιράκ. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η συζήτηση, θα προχωρήσει περαιτέρω και προβλέπεται μια σημαντική συνάντηση στη Σαουδική Αραβία για το θέμα αυτό. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Δεν είναι μονάχα στρατιωτικό θέμα αυτό, έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση αυτή τη ομάδα, έχει να κάνει με την παρουσία ξένων μαχητών, που είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τι δυνάμει τη ε, υπηρεσία πληροφοριών μα. Έχει να κάνει και με την αντιμετώπιση τη ιδεολογία που υποστηρίζει αυτό το κίνημα και δεν έχει να κάνει με άμεση στρατιωτική παρέμβαση από εμά, αλλά για υποστήριξη με αυτού που αντιμετωπίζουν το μόρφωμα αυτό Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει μια πιο συντονισμένη προσπάθεια μέσα στην οποία το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να παίξει ένα περιορισμένο ρόλο. Ένα τρίτο σύντημα τώρα, οι ανοιχτέ πύλες του ΝΑΤΟ, αυτό το συζητήσαμε. Υπήρξε και πάλι μια επαναεπιβεβαίωση αυτής της πολιτικής ανοιχτών θυρών. Όπως ξέρετε η Γεωργία είναι μια χώρα η οποία έχει ε, την θέληση να προχωρήσει προς μια μεγαλύτερη προσέγγιση με τον ΝΑΤΟ και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα να ενισχύσει την ε, αμυντική της ικανότητα. Έχουμε προχωρήσει σε πιο πολύ σε βάθος συνομιλίες με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για να αντιμετωπίσουμε τα εκρεμή θέματα <clears throat> ώστε να προχωρήσουμε στο τέλος του 2015 σε μια συνάντηση σε επίπεδο ε, υπουργικό ώστε να μπορέσει να απευθυνθεί ενδεχομένως πρόκειται για το Μαυροβούνιο, μια πρόσκληση στη χώρα αυτή να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν παροτρινθεί από την πολιτική μας ανοιχτών θυρών και αυτό θα ενισχύσει τη σταθερότητα η οποία βοηθά την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Για τις εταιρικές σχέσεις πήραμε δύο κέρδιες αποφάσεις. Καταρχήν να φτιάξουμε μια πλατφόρμα διαλειτουργικότητας. Αυτό είναι τεχνικό βέβαια, αλλά αυτό σημαίνει ότι μαζί με, τις, ε, με τους επιχειρησιακούς μας εταίρους έχουμε δημιουργήσει ένα επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των στρατιωτικών δυνάμεών μας, δηλαδή ξέρουν πώς να συνεργαστούν σε τεχνικό επίπεδο τα συστήματα δίκησης και ελέγχου, οι επικοινωνίες, οι υπολογιστές, όλα αυτά ξέρουν πώς μπορούν να συνδεθούν οι στρατιωτικές δυνάμεις όταν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό έχει φτάσει ένα πρωτοφανέ επίπεδο. Ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε τόσο μεγάλο επίπεδο ολοκλήρωση, τουλάχιστον δυνητική ολοκλήρωση μεταξύ τόσων πολλών στα, ε, ενόπλων δυνάμεων μέχρι ενό επίπεδου μικρών μονάδων. Αυτό είναι λοιπόν ένα μεγάλο ατού για τι επιχειρήσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του, του ΟΗΕ αλλά και του ΝΑΤΟ τα πρότυπα του ΝΑΤΟ γίνονται όλο και περισσότερο τα διεθνή πρότυπα και υιοθετούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι θετικό για όλου. Επομένω, έχουμε δημιουργήσει αυτή τη δομή να βοηθήσει την περαιτέρω ολοκλήρωση. Δεύτερον, έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα βελτιωμένων ευκαιριών, το οποίο σημαίνει ότι οι χώρε οι οποίε είναι πιο προχωρημένε, έχουν τη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, είναι πιο δεσμευμένε για μια εταιρική σχέση με τον ΝΑΤΟ, θα μπορούν να έχουν πιο έντονο πολιτικό διάλογο και πιο έντονη ενσωμάτωση στις δομές του ΝΑΤΟ και την οργάνωση του ΝΑΤΟ και στις ασκήσεις κτλ. Διεθνείς οργανισμοί τώρα. Είχαμε την πρώτη συνάντηση των Υπουργών με την ε, ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης και φυσικά ήταν παρόν ο κύριος και η Άστον και σε αυτές τις συναντήσεις. Και με τον τρόπο αυτό τονίζω αυτά τα οποία είπα και προηγουμένω χρειάζεται να έχουμε καλύτερο συντονισμό, καλύτερη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων. Έχουμε φυσικά πολύ καλή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την ΟΑΣΕ όταν αυτό <clears throat> απαιτείται. Με το Συμβούλιο της Ευρώπης βέβαια έχουμε λιγότερες σχέσεις. Θέλουμε λοιπόν να βελτιωθεί και αυτή η συνεργασία και το αναφέρει και το τελικό μας ανακοινωθέν. Και τέλος, προσπαθώ και εδώ να είμαι σύντομος, Αφήνω κατά μέρος αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως. Ήθελα να σας πω ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει διορίσει ένα ειδικό εισηγητή για την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες σε ένοπλες ζώνες και την ασφάλειά τους. Αυτό είναι μια ειδική θέση και καταδεικνύει και την ε, θέληση που έχει το ΝΑΤΟ να παίξει ένα ειδικό ρόλο στον τομέα αυτό. Ένα παράδειγμα. Πολλά από τα θέματα που εμπίπτουν στο ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας, έχουν ενσωματωθεί στην εκπαίδευση που δίνουμε στους ε, στρατιωτικούς. Υπάρχουν εκατομμύρια στρατιωτικών τώρα που έχουν την εκπαίδευσή τους να προσαρμόζεται να σέβονται λοιπόν αυτό το ψήφισμα και να εξασφαλίζουν ότι η προστασία των γυναικών σε ενοπλες είναι τμήμα της ε, Εκπαίδευση τους. Και νομίζω ότι μπορώ σε αυτό το σημείο να σταματήσω. Ευχαριστώ κύριε Αναπληρωτή. Βοηθάει Γενικό Γραμματέα. Άρχισε η συζήτηση. Αποσία του κυρίου Γκάλερ. Τι αποσία, εδώ είμαι. Ε, εντάξει. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Όχι, όχι. Δεν ζήτησα το λόγο. Ε, άκουσα, δεν έχω συγκεκριμένη ερώτηση επικαιρή ε, να κάνω. Ο κύριος Παρνιό τότε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η επισκόπηση αυτή της κατάστασης από πλευράς ΝΑΤΟ είναι ακριβής όσο και ενδιαφέρουσα αλλά και άκρο σημαντική. Έχω μια ερώτηση, μάλλον παρατήρηση να σας κάνω. καλά το είπατε. Έχουμε πολλές αποστολές με το ΝΑΤΟ και γενικότερα με όλες αυτές τις χώρες που τώρα κάνουν πόλεμο κατά αυτών των δολοφόνων και τρομοκρατών. Και δεν θα πρέπει να τους ε, ε αναδεικνύουμε και να τους χαρακτηρίζουμε κράτος, Ισλαμικό κράτος. Είδαμε και το μεγάλο μουφτή της Αιγύπτου που καταδικάζει σήμερα και λέει κυρίως να μην ε, συγχέουμε τις έννοιες και να μην πούμε ότι πρόκειται για κράτος που ε, θα έρθει να αντικαταστήσει ένα άλλο η καταπολέμηση αυτής της ιδεολογίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο και σημαντικό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να μπορέσουν να μπουν στη Μεγάλη Συμμαχία και στο συνασπισμό αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε δράση. Γιατί αυτοί οι τρομοκράτες αυτοποκαλούνται Σουνίτες μουσουλμάνοι Οπότε μπορεί να υπάρχει μια πολιτική και ιδεολογική προσέγγιση με τη συμμετοχή ε, των Εμμυράτων. Σε ό,τι αφορά τους ξένους μαχητές, έχετε δίκιο. Και εκεί οι υπηρεσίες προφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να παίξουν το ρόλο τους για τη δράση στην επικράτειά μας. Είδαμε πολύ πρόσφατα τι έγινε στη Γαλλία και το άλλο σημείο να κοπεί η χρηματοδότησή τους υπάρχει δυσκολία βλέπουμε γιατί αυτή η τρομοκρατική ομάδα έχει μια χρηματοδότηση και ήταν αφετηρία για την εισβολή εκεί στο Ιράκ. Δεν είναι μόνο, έχουν και εξωτερική χρηματοδότηση και είναι πολύ σημαντικό να φέρουμε κοντά μας και τη Σαουδική Αραβία που όπως ξέρουμε δυστυχώς ήταν και αυτή η πηγή χρηματοδότησης ε, αυτού που αυτοποκαλείται τώρα και χαλιφάτο. Σας ευχαριστώ. Οι συντονιστέ δικαιούνται πρώτα να λάβουν το λόγο. Ο κύριο Μάρεκ Γιούρεκ, εκ μέρου των μεταρρυθμιστών συντηρητικό, θέλει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Στην πρώτη μου ε, ομιλία περιορίστηκα στην Ουκρανία. Τώρα θα επανέλθω πάλι στην Ευρώπη, γιατί μιλήσατε για την διεύρυνση της συμμαχίας στην Ευρώπη με το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνιο και άλλες χώρες. Πιστεύω όμως ότι για τη γενική ασφάλεια της Ευρώπης, όχι μόνο για τις Βαλτικές χώρες και την Πολωνία ή τις χώρες των Ανατολικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ πιο σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη τώρα είναι οι διαπραγματεύσεις και η πιθανή πρόσκληση της Γεωργίας στην Ευρωατλαντική Συμμαχία αντί να προσκαλέσουμε το Μοντενέγκρο το Μαυροβούνιο γιατί μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας νομίζω ότι μια αντίστοιχη και συμμετρική αντίδραση ήταν η πρόσκληση της Γεωργίας και έχουμε και το θέμα της Ουκρανίας και της τελευταία τον τελευταίο χρόνο ακούγεται, το... την πρόταση... ακούγεται η πρόταση για την ένταξη της Ουκρανίας, αλλά για την ε, Γεωργία υπήρχε συμφωνία σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των, ε, των βλέψεων της Γεωργίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι τόσο επίμαχο το θέμα. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να χάσουμε χρόνο στη συζήτηση των νομικών λεπτομεριών της ένταξης της Γεωργίας, αλλά να ε, καταρτήσουμε έναν οδικό χάρτη για μία όχι πολύ σε, μεταγενέστερο χρόνο, σχετικά σύντομα ε, ένταξη της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Γιατί πιστεύω ότι χωρί διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να ικανοποιήσουμε ένα λαό που θέλει να γίνει σύμμαχός μας. Κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μερικές ερωτήσεις για το Αφγανιστάν. Παρακαλώ να κάνω. Στην Οαλία δηλώσανε για το Αφγανιστάν και παραθέτω έχουν γίνει μεγάλες προόδοι στην παιδεία, την υγεία, την οικονομική ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αμελιώδεις ελευθερίες, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Τέλος της παράθεσης. Μα είναι πιστευτά αυτά τα πράγματα, 7,4 εκατομμύρια από τα 26 εκατομμύρια κατοίκων ε, ε, είναι περίπου ε, σε λοιμό και ακόμα 8 εκατομμύρια υποσυτίζονται, 27% του πληθυσμού έχουν πρόσβαση ε, σε πόσιμο νερό. Μόλις 5% σε ε, εγκαταστάσεις υγιεινής ε, κτλ. Τώρα είναι πιστευτό πραγματικά ότι έχει βελτιωθεί τόσο πολύ η κατάσταση. Υποτίθεται. Άλλη ερώτηση. Διμερή συμφωνία ασφαλείας, διμερή συμφωνία ασφαλείας είναι η προϋπόθεση ε, για την ε, ε, αποστολή που θα διαδεχθεί το ΝΑΤΟ, Resolute Support. Δεν υπάρχει μια τέτοια διμερή συμφωνία όμως. Και τι θα γίνει, θα αποχωρήσουν όλα τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ και με την επιμελητία, τι γίνεται, ακόμα 40.000 εκεί τα στρατεύματα στο Αφγανιστάν, είναι φυκτά αυτά τα πράγματα. Άλλη ερώτηση. Το Resolute Support θα υποστηρίζει και άμεσα επιθέσεις των ε, αφγανικών ενόπλων δυνάμεων. Και σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν εδώ, κοστίζουν 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και εξασφαλίζεται χρηματοδότηση μέχρι το 2017. Θεωρείτε ότι η Δύση και μετά θα πληρώνει τη μερίδα του λέοντος. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Ο αφγανικός προπολογισμό θα είναι σε θέση να υποστηρίζει τέτοια ποσά. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Mrs. Sorry. Ευχαριστώ κυρία Σεμπάη. Σας λέω όλο κύριο, λυπάμαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ενδιαφέροντα αυτά που ακούμε. Ότι δεν υπάρχει συμφωνία ε, γραπτή και επίσημη για διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ε, γιατί άλλα ακούμε. Ε, αλλά είτε έχει γίνει γραπτός αυτό είτε προφορικά, έχει δεσμευτεί προς τη Ρωσία το ΝΑΤΟ να μην διευρυνθεί προς Ανατολάς. Είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί. Επίσης η Ρωσία συχνά παραβιάζει μεν τις συμφωνίες, εμείς δεν τις παραβιάζουμε τις ίδιες μας συμφωνίες με τη Ρωσία. Ας πούμε τη συμφωνία ΝΑΤΟ-Ρωσίας, όπου λέγουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνεργασία ε, και ε, και στο εσωτερικό μας ε, ε, θα πρέπει να στραφούμε περισσότερο προς τη διαλειτουργικότητα και τη συμβατότητα των όπλων δυνάμεων αντί συνεχώς να σταθμεύουν δυνάμεις μας σε προκεχωρημένα φυλάκια όλο και πιο μακριά. Στη Βαλτική, στη Ρουμανία, στην Πολωνία, τι δυνάμεις θα αναπτυχθούν. Και έχω και μια ερώτηση για την αποστολή στο Αφγανιστάν, η Νίσαφ. Επανειλημμένα έχω μεταβεί προσωπικά στο Αφγανιστάν και επισκέφθηκα ε, τους Σουηδούς που σταθμεύουν εκεί και τους Γερμανούς και ήμουνα και στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ εκεί και τότε ήμουν μέλος της Σουηδικής Βουλής και ε, ασχολούμουν και με την πολιτική υποστήριξη προς το Αφγανιστάν, όχι τη στρατιωτική. Και εκεί είδα και συναντήθηκα με πολλούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα και στην τελευταία μου επίσκεψη στο Αφγανιστάν ήταν ξεκάθαρη εικόνα ότι έλεγε ο κόσμος ότι πρέπει να φύγουν τα ξένα στρατεύματα. Γιατί είναι αδιέξοδη η ε, πολιτική που ακολουθούμε. Και ρωτώ, έχει αλλάξει η κατάσταση. Έχει επηρεαστεί η κατάσταση από το Ιράκ, έχει αλλάξει η στάση ε, των Αφγανών ε, αμάχων ε, ως προς την παρουσία ξένων στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. Αυτά ευχαριστώ. Thank you. Mr. Κύριε Έλερ, θέλετε να λάβετε εσείς το λόγο. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε αυτό που αναφέρατε σε σχέση με τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, γιατί ορισμένοι από εμά ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, αλλά και για τους προϋπολογισμούς. Αυτό που μάθαμε από το παρελθόν ήταν ότι αυτή η συνεργασία ήταν πολιτικά επιθυμητή, αλλά σε πρακτικό επίπεδο δεν έλαβε ουσιαστικά χώρα και δεν είχε χρηματοδότηση. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι το εξής. Μήπως μπορεί να υπάρξει πιο συγκεκριμένη αναφορά για συγκεκριμένα σχέδια και σε τι σχέδια συνεργασίας και αντίθετα, αντίστοφα από τη δική μας πλευρά, εμείς έχουμε προετοιμάσει προϋπολογισμό για μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της ε, ασφάλειας, ιδίως των ε, πληροφοριών. Και επίσης έχουμε αναφερθεί στην ενδιάμεση ε, λύση για αερομεταφορά που έχει να κάνει με τις δυνάμεις ταχείας αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν επίσης πιο λεπτά θέματα όπως είναι η συνεργασία πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων. Υπήρξε μια εκπαίδευση η οποία έγινε στο ΝΑΤΟ πριν από μερικά χρόνια χωρίς να λαμβάνεται υπόψη καθόλου η παρουσία της Ευρώπης και οι ικανότητες της να συμβάλλει στην αντιμετώπιση πολιτικών κρίσεων ενώ στην πράξη οι δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίζουν σημαντικό ρόλο σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τα τρία αυτά θέματα αντιμετωπίστηκαν πέρσι σε επίπεδο προπολογισμού. Θα ήθελα να ξέρω αν σε πολιτικό επίπεδο υπήρξε από την πλευρά του ΝΑΤΟ κάποια σκέψη για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ για τον ε, Ραντός από το Άλντε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. στην δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ουαλίας. Οι αρχοί κρατών συμφώνησαν ότι το σχέδιο δράση για την ετοιμότητα θα εγκριθεί και μάλιστα κοινέ ομάδε κρούση υψηλή ετοιμότητα προβλέπονται που θα είναι αναπτυξίμες μέσα σε λίγες μέρες. Αυτές οι κοινέ ε, ομάδες κρούσης ε, υψηλής ετοιμότητας είναι τμήμα των ε, ομάδων αντίδρασης του ΝΑΤΟ και μοιάζουν με, τις, με τους μάχημους σχηματισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, πριν από δύο μέρες, οι Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίασαν στο Μιλάνο με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάσκεψή τους τις Ευρωπαϊκές Μάχημες Μονάδες, τα Battle Groups. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά κατά νου, θα ήθελα να σας υποβάλω δύο ερωτήσεις, κυρία Πατουράη. Η πρώτη ερώτηση είναι γενική. Πώς και πότε θα σχηματιστούν αυτές οι ομάδες ε, ε, κρούσεις ε, ύψης της ετοιμότητας, γιατί στη, η δήλωση, η διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής της Ουαλίας λέει ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσεως ετοιμότητας θα ξεκινήσει πάρα αυτά, αμελητή. Δηλαδή, η διαδικασία ήδη ξεκινά. Και δεύτερη ερώτηση, πιο σημαντική από την άποψη των δικών μας ενδιαφερόντων της Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ. Οι μάχημες ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά τα battle groups της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λάβουν μέρος στην, στις κοινέ αυτές ομάδες κρούσης υψηλή ετοιμότητας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καστάλντο. Μία ερώτηση για το Αφγανιστάν. Μιλήσατε για 46 δις, ε, ε, δεν ξέρω αν ήταν ευρώ ή δολάρια για τις δυνάμεις του Αφγανιστάν. Ε, τεράστιο ποσό. Τι έλεγχος γίνεται για τη χρήση των κονδυλίων αυτών και τι κινδύνους έχει μια τέτοια χρηματοδότηση. Γιατί έχουμε πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις στο Αφγανιστάν. Ας μην ξεχνούμε τι συνέβη στο Ιράκ. Τώρα, για το Ιράκ και το αυτοαποκολούμενο Ισλαμικό κράτος. Η αποστολή βοήθειας στο Ιράκ που μας είπατε, ε, πότε θα δοθεί ε, μετά τη σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ή θα πρόκειται για μια αποστολή που θα δοθεί στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Ευχαριστώ κυρία Άννα Σας ευχαριστώ. Πρόσφατα ακούσαμε τον πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βαγδάτη που μας είπε ότι μερικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν στρατητικό εξοπλισμό σε ε, Ιρακινούς, ιδιαίτερα στο Κουρδιστάν και η παροχή αυτών των εξοπλισμών είναι τελείως εκτός ελέγχου. Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουν, ποιοι θα είναι οι τελικοί παραλήπτες. Αυτό ανησυχεί, προβληματίζει τον Άτομο μια τέτοια κατάσταση. Επίσης, ο κύριος Ποπόφσκι μας μίλησε νωρίτερα για τη Λιβύη και είπε ότι και η Λιβύη απασχολεί ιδιαίτερως ε, τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Φαντάζομαι και τους ε, συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Ε, πέραν των προβληματισμών και παίρνουν το ότι έχουμε τη Λιβύη στο μυαλό μα. Έχουμε κάτι πιο απτό, κάτι στα χέρια μας, καμιά πρωτοβουλία συγκεκριμένη, κάποια συντονισμένη πρωτοβουλία με τους ε, Άραβες γειτονέ μας, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κόουζου. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση για το Ιράκ. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και την ιστορία όμως, το ιστορικό έγιναν μία, έγινε μία τσαπατσούλικη προσπάθεια ε, μετά από μια παράνομη εισβολή. Γι' αυτό είναι σημαντικέ οι αποδείξει. Με καταστροφή των εθνικών ε, δομών του Ιρακινού κράτου ε, με, με τρομερή εισβολή και με τη διαφορά μεταξύ των φατριών και επίσης την υποστήριξη των Μαλίκη και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι και σύμμαχος του Ιράν. Τώρα, κύριε Ιπατουράη, ποια θα είναι η σχέση αυτής της αποστολής με τον ΟΗΕ. Θα ζητήσουμε εντολή από τον ΟΗΕ ή είναι ένα ακόμη ένα βήμα να υποκαταστήσει τον ΝΑΤΟ τον ΟΗΕ. Επίσης, τις συναντήσεις που έχετε με τη Σαουδική Αραβία θα ζητήσετε ε, στοιχεία για τις αποδείξεις ε, ή ε, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση σε τρομοκρατικές οργανώσεις ε, ή μήπως θα συνεχίσει η Σαουδική Αραβία να κάνει ό,τι θέλει. Ο κύριος Συναδεινός. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω αυτό που είχα ξεκινήσει και διακόπηκε και αφορά την προσφώνηση του Υπουργού της Φύρομ στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουαλία ως Υπουργού της Μακεδονίας. Πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι έγινε εκ παραδρομής και όχι εσκεμένα. Περιτώ βέβαια να σας θυμίσω ότι η συμμαχία της οποίας είμαστε μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία της Ευρώπης, αλλά και πλήθος άλλων θεσμικών οργάνων, αναφέρονται σε αυτή σύμφωνα με τις αποφάσεις 817 και 845 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Όπως επίσης είναι περιττό να θυμίσω ότι η Συμμαχία στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008 αποφάσισε την αναβολή της πρόσκλησης ένταξης της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ εφόσον δεν λυθεί το ζήτημα της ονομασίας. Ρωτώ λοιπόν αν υπάρχει λιμένη απόφαση από το ΝΑΤΟ ερήμην των μελών του για την αποδοχή της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ ως Δημοκρατία της Μακεδονίας και απλά είναι θέμα χρόνου και όχι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Γνωρίζετε επίσης ότι η Μακεδονία εδώ και 4-5 χρόνια αναφέρεται στην ελληνική ιστορία ενώ το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια για τη Φύρομ αναφέρεται από το 1945. Αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός δεν σέβεται κατά την άποψή μου την ιστορία των κρατών μελών του. Επίσης σαν αντιπαραβολή θα ήθελα να σας θυμίσω τη διένεξη της Γαλλίας με τη Βρετανία για την είσοδο της Μεγάλης Βρετανίας το 1970 και κάνω έναν παραλληλισμό γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Oh, Ευχαριστώ, ο Δούδα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αναπληρωτή Γενική Γραμματέα, υπάρχει κάποιος χριστιανικός σύνδεσμος στο Ιράκ. Είσαστε έτοιμοι ή εξετάζετε τη δυνατότητα να προστατεύσετε αυτό τον οργανισμό, αυτή την ένωση. Σας ευχαριστώ. Έχουμε κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών και θα ήθελα τώρα... Α, συγγνώμη. Κύριε Σαφχάουζεν, παρακαλώ σύντομα. Εγώ θέλω να ακολουθήσω αυτό που είπε ο συναδελφός μου στο Ιράκ, στη Συρία και στη Λιβύη, στις χώρες αυτές όπου έχουμε παρέμβει υπάρχει μια τάση να εξοντωθούν οι χριστιανοί. Τι θα κάνετε για να αποτρέψετε αυτή την κίνηση που γίνεται και ιδίως σε σχέση με όλα αυτά τα ένοπλα στοιχεία τα οποία έχουν αποφασίσει να εκδιώξουν ή να εξαλείψουν τους χριστιανούς από τη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ κύριε Απατουρά, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω διαδοχικά όλα αυτά τα στοιχεία. Εγώ συμμεριζόμαι απόλυτα την ε, ανάλυση ότι το να αντιμετωπίσουμε την ιδεολογία των τσιγαντιστών απαιτεί και την υποστήριξη των ε, Αραβικών Εμμυράτων και η Σαουδική Αραβία θα πρέπει και αυτή να παίξει κάποιο ρόλο στη χρηματοδότηση αυτής της προσπάθειας. Το γνωρίζει αυτό η Σαουδική Αραβία, γι' αυτό στη Τζέντα θα είναι οικοδεσπότες μια συνδιάσκεψης. Αλλά ξέρουμε ότι η Σαουδική Αραβία είναι και η χώρα που έχει τις πιο σημαντικές ιερές τοποθεσίες του Ισλάμ και γι' αυτό έχει μεγάλη αξιοπιστία. Και αν ενισχύσουν τον αγώνα τους κατά της ακραίας ιδεολογίας, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται. Συμμερίζομαι λοιπόν την ανάλυση της σας. Για τη γεωργία και τυχαίνει να είμαι ο ειδικό εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ για τον Κάφκασο και την Κεντρική Ασία και έχω περάσει πολύ καιρό στην ε, Γεωργία προσπαθώντας να σας βοηθήσω να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι μια πολιτική του ΝΑΤΟ και μια απόφαση έχει ληφθεί ότι θα γίνουν μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλω αυτό να γίνει το ταχύτερο δυνατό όπως θέλουν και όλοι οι σύμμαχοι μας του ΝΑΤΟ. Η δέσμη αυτή μέτρων η οποία ενεκρίθη στη διάσκεψη κορυφής είχε σαν στόχο να ενισχύσει τους, τους γεωργιανούς να ενισχύσουν την ε, στρατηγική τους ικανότητα, να υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του ΝΑΤΟ, <clears throat> μεγαλύτερη συμμετοχή σε κοινέ ασκήσεις, περισσότερες διευκολύνσεις του ΝΑΤΟ στην Γεωργία, μεγαλύτερη συμμετοχή της Γεωργίας σε στρατηγικέ συζητήσεις για τις δυνάμεις αντίδρασης του ΝΑΤΟ, σε ασκήσεις, σε σχολεία. Θα υπάρξουν λοιπόν και θα υπάρχει μεγαλύτερη παρουσία του ΝΑΤΟ στα Υπουργεία του, της Γεωργίας για να τους βοηθήσουμε να ενισχύσουν την παρουσία τους μέσα στο ΝΑΤΟ όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας των Πρόεδρων της Ιωρίας, όλα αυτά είναι ουσιαστικά, δεν είναι ευχολόγια, δεν είναι λόγια μονάχα, δεν είναι ίσως αυτά που θέλουν όλοι να ακούσουν, αλλά είναι πάρα πολύ θετικά και μας ικανοποιούν ιδιαίτερα. Και θα συμμετάσχουμε στην εφαρμογή όλων αυτών. Για το Αφγανιστάν. Εγώ απασχολούμαι με το Αφγανιστάν για πάρα πολλά χρόνια. και έχω πάει πολλές φορές μέσα στο 2014 και είναι πάρα πολύ σαφή τα στοιχεία που δείχνουν ότι έχει βελτιωθεί η ζωή του μέσου Αφγανού. Ένα τέτοιο στοιχείο λοιπόν είναι το ότι όταν η διεθνής κοινότητα μπήκε στο Αφγανιστάν το 2001 το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης για ένα Αφγανό ήταν περίπου 36 χρόνια. Αυτή ήταν τότε η κατάσταση. Σήμερα είναι περίπου 56 χρόνια το προσδόκιμο επιβίωση. Σε αυτό το λοιπόν σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε βελτιώσει την ε, προσδοκία ζωής για τους Αφγανούς. Πολλοί Αφγανοί λοιπόν ζουν <clears throat> οι οποίοι δεν θα ζούσαν χωρίς την διεθνή προσπάθεια και την στρατιωτική παρουσία. Όλα αυτά λοιπόν τα έχετε δει και τα έχει δει και η Σουηδή συνάδελφός μας. Έχει βελτιωθεί η προστασία των ε, ε, βρεφών και των μητέρων έχουν μειωθεί οι αντίστοιχε νησιμότητες και ήμουνα παρόν σε μια συνάντηση με την επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας του Κοινοβουλίου της, ε, του Αφγανιστάν που είναι γυναίκα. Αν λοιπόν είναι γυναίκα αυτή η οποία ασχολείται με τα θέματα αυτά και είναι κάτω από 40 ετών Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία είναι πάρα πολύ θετικά και καταδεικνύουν πόσα θετικά πράγματα έχουν γίνει στο Αφγανιστάν χάρη στην παρουσία της διεθνούς αυτής δυνάμεως και φυσικά εκφράσουν και αυτοί την ευγνωμοσύνη τους. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα, της, ε, στο θέμα αυτό της διεθνούς παρουσίας. Έχετε δίκιο, είναι πολλοί Αφγανοί οι οποίοι δεν θέλουν να συνεχιστούν οι ένοπλες συγκρούσεις στο χώρο τους. Και το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Και φτάνει πάντα ένα σημείο, δεν λέω ότι αυτή τη στιγμή θα ισχύσει αυτό, όπου η διεθνής παρουσία δεν είναι πια ε, θετική, δεν βοηθάει πια. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά οι, Αφγανιστές, οι αφγανικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να αναλάβουν όλο αυτό τον αγώνα. Εμείς έχουμε επενδύσει δισεκατομμύρια στο να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με επαρκή εκπαίδευση και χρηματοδότηση και παροχή συμβουλών μπορούν να συνεχίσουν οι ίδιοι την ε, αντιμετώπιση σε στρατιωτικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλές βέβαια δυσκολίες, αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν πια ασφαλή καταφύγια για τους τρομοκράτες στο Αφγανιστάν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό όπου μπορούμε να τους παραδώσουμε τη σκητάλη και το ΝΑΤΟ λοιπόν δεν θα έχει πια ρόλο ε, ε, μάχημο στην περιοχή. Δεν θα έχουμε δυνάμεις οι οποίες θα βρίσκονται επιτοπίως, θα έχουμε φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε επίπεδο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων <clears throat> και δεν θα υπάρχει μάχημη παρουσία στο Αφγανιστάν από την 31η Δεκεμβρίου του 2014. Τώρα, αν υπάρχει δυνατότητα σε επίπεδο επιμελητίας να αποσύρουμε τις δυνάμεις μας, δεν ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και τι θα κάνουμε όταν σταματήσει η παρουσία μας, Δεν είμαι πιο σαφής. Δεν ε, είπα 46 δισεκατομμύρια δολάρια, ήταν, είπα από 4 μέχρι 6 δισεκατομμύρια, όχι 46, 4 μιλάω πάρα πολύ γρήγορα. Ε, ήταν τεράστιο φυσικά το άλλο ποσό. Ε, και θα δούμε από εκεί και πέρα. Ελπίζουμε η αφγανική οικονομία να έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορέσει να υπομειστεί το μεγαλύτερο βάρος αν χρειαστεί όμως και περαιτέρω υποστήριξη μετά, ε, είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά ένα βήμα κάθε φορά ε, για τα επόμενα έτη είναι επαρκής η χρηματοδότηση και είναι εντάξει. Για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Ο συνάδελφος Άλεξ ε, Πατριάνου είναι πάρα πολύ ειδικό. Θα σας δώσω το νούμερό του να το πάρετε τηλέφωνο για να συζητήσετε όλα αυτά τα θέματα ε, είναι μεγάλα και μικρότερα ε, τα έργα και οι τομείς συνεργασίες, όπως ε, ξέρετε ο αναπληρωτής γενικός διοικητής των δυνάμεών μας είναι και διοικητής των ευρωπαϊκών δυνάμεων και ο Οργανισμός ε, Άμυνα Ευρωπαϊκός συνεργάζεται στενά με τις δικές μας δομές για να μην υπάρχουν επικαλύψεις. Αλλά υπάρχουν κάποιες πολιτικές συζητήσεις, κάποια έγγραφα που είναι πολύ δύσκολο να συνενώνονται πάντα για να συζητούν από κοινού. Ε, είναι θέματα επιτελείων. Για περισσότερες λεπτομέρειες σας παραπέμπω στον συνάδελφό μου με χαρά να σας τα πει. Τώρα, για την επαναβεβαίωση και για την εχμή του δόρατος. Έχει ήδη αρχίσει η εφαρμογή. Ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, που είναι υψηλό βαθμός ανώτατος αξιωματικός, εχθές στο Συμβούλιο μίλησε στους πρέσβεις και είπε «Ξέρουμε τι θέλουμε και ξέρουμε ο καθένας από σας τι έχει ως δυνατότητες και θα έρθουμε σε εσά για να πάρουμε ό,τι μας χρειάζεται». Και η βασική προσέγγιση αυτής της γενιάς δεν είναι να περιμένεις ο καθένας να σου δώσει ό,τι μπορεί. Είναι περίπλοκος αυτός ο μηχανισμός. Θα πρέπει ο καθένας να δίνει το σωστό εξάρτημα για να υπάρχει η σωστή συνεργασία. Ήδη έχει αρχίσει αυτή η προσπάθεια με τις εθνικές κυβερνήσεις για να έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι πολλές κυβερνήσεις ήδη έχουν δηλώσει εθελοντικά πολύ ειδικέ δυνατότητες που χορηγούν. Έχει αρχίσει λοιπόν ήδη αυτή η διαδικασία και μπορώ να σας διαβεβαίσω ότι Καταλήγοντας, ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι ελπίζει αυτό να γίνει όντως αμέλητη. Σε ύψιστο επίπεδο θα γίνει η παρακολούθηση και η συνέχεια. Δεν νομίζω ότι οι μάχημοι σχηματισμοί έχουν σχέση με αυτό. Καμία σχέση. Μπορεί να σπάλω, αλλά δεν είναι, κάτι διαφορετικό. Τώρα, για την υποστήριξη στο Ιράκ. Εξ όσων γνωρίζω, δεν είναι το ΝΑΤΟ αλλά εξ όσων γνωρίζω, θα πάει και στις ε, δυνάμεις ασφαλείας ε, του Ιράκ, τις Ιρακινές ενόπλες δυνάμεις και στους Κούρδους Πεσμεργά. Ήδη συμβαίνει αυτό ε, στους Κούρδους μαχητές για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πέσουν σε λάθος χέρια τα όπλα. Ξέρουμε όμως όταν κατέλαβε κάποιο έδαφος αυτή η τρομοκρατική ομάδα έφτασαν στα χέρια της περίπλοκα όπλα και συστήματα που γαρονικά δεν θα έπρεπε και κανείς δεν το επιθυμεί αυτό για τη Λιβύη. Είναι μια πάρα πολύ ατυχής κατάσταση για όλους και μεταξύ αυτών για χώρες που δέχονται τόσους πολλούς παράνομους μετανάστες. Προσωπικά έχω μεταβεί στη Λιβύη στην περίοδο μετά τη στρατιωτική επιχείρηση και τον τερματισμό της κατόπιν αιτήματος των Λιβικών αρχών μας ζήτησαν να τους βοηθήσουμε να στηθεί το Υπουργείο Αμήνης, η Πολιτική Ασφαλείας και να τους δείξουμε πώς διοικείς μια τέτοια δομή ως χώρα δεχθήκαμε αυτή την αίτηση, το αίτημά τους και πήγαμε. Ήμασταν έτοιμοι. Αλλά η κατάσταση επιδεινώθηκε πάρα πολύ, η κατάσταση ασφαλείας, όπως γνωρίζετε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη ε, γνωρίζουν τεράστιες δυσκολίες και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρουμε ποιος είναι η κυβέρνηση να απευθυνθούμε. Από ό,τι φαίνεται είναι δύο κυβερνήσεις και διάφορες ε, πολιτοφυλακές και το περιβάλλον ασφαλείας είναι πάρα πολύ ε, περίπλοκο. Έχει παγώσει κάπως αυτή η προσπάθεια, αλλά αν υπάρξει ασφάλεια και μας καλέσουν, ε, είμαστε πρόθυμοι να πάμε. Και τι πρέπει να γίνει ξέρουμε και πώς να το κάνουμε ξέρουμε σε στενή συνεργασία με τους ε, συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Για μένα ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό αυτό το παράδειγμα. Παρά όλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε καμιά φορά για πολιτικούς λόγους, ε, ε, στις έδρες και στα αρχηγεία ε, όταν φτάνεις επί τόπου και χρειάζεται να συνεργαστείς για την ζωτική σημασία όλα δουλεύουν και στο Κόσοβο και στο Αφγανιστάν και αλλού και παντού. Για το Ιράκ και την εντολή. Δεν ξέρω τι θα κάνει το ΝΑΤΟ, αν κάνει οτιδήποτε το ΝΑΤΟ, αλλά Έχουμε ένα ε, συμπεφωνημένο διμερές πλαίσιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τις συμφωνίες συνεργασίας και αν προσκληθεί το ΝΑΤΟ δεν χρειάζεται εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας. Κατά τα άλλα είναι πολύ ισχυρά τα ψηφίσματα έτσι και αλλιώς του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανάγκη καταπολέμηση αυτής της απειλής, αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης και δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε νέα εντολή αυτό είναι κάτι που βρίσκει σύμφωνη όλη τη διεθνή κοινότητα. Τώρα, είχαμε την ερώτηση για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και το όνομα. Ε, η θέση μας για το όνομα είναι σαφής. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις και δεν κάνω εγώ τις ανακοινώσεις βέβαια, ειλικρινά. Αν υπήρξαν ασφάλματα, ε, ήταν ασφάλμα αυτό, ε, είναι γνωστή η θέση μας. Για τις χριστιανικές κοινότητες, νομίζω υπάρχει μεγάλη ανησυχία γενική στις χώρες ΝΑΤΟ για όλες τις κοινότητες και τους χριστιανούς, αλλά όχι μόνο τους χριστιανούς. Είναι ακραία η βία και οι ομότητες εκεί στην περιοχή με στόχο κυρίως άλλους μουσουλμάνους και διάφορες αιρέσεις και είναι πολλές οι αιρέσεις εκεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό χωρίς να παραμελούμε τους χριστιανούς αλλά σκεφτόμαστε και τους άλλους ε, που σκοτώνονται και να μην θεωρούμε ότι είναι ας πούμε ε, ίσονο σημασία έχει λιγότερη αξία η ζωή τους επειδή δεν είναι χριστιανοί. Όλες τις θρησκευτικέ ε, και εθνικές μειονότητες, αιρέσεις και ομάδες αξίζουν την ίδια προσοχή από πλευράς μας και φροντίδα και ελπίζω να τους δοθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πατουράη. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο παραπάνω ε, σε αυτό το πλαίσιο, τη συμφωνίες πλαίσιο, δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Αν άκουγε ένας Πολωνός δεν θα καταλάβαινε πάρα πολύ τι εννοείται, θα μπορούσατε λίγο να το εξηγήσετε. Η ιδέα αυτή της, ε, του πλαισίου είναι σαν τη μάχη με ομάδες, αλλά δεν πρόκειται για στρατιωτική ανάπτυξη. Όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ έχουμε και μεγάλες χώρες με μεγάλες στρατηγικές ικανότητες και ικανότητες πλήρους φάσματος και έχουμε και μικρότερες χώρες με χαμηλότερους αμυντικούς προϋπολογισμούς και δεν ε, έχουν ε, ε, ένοπλες δυνάμεις πλήρους φάσματος ούτε μπορούν να αναπτύξουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες γιατί κάτι τέτοιο είναι δαπανηρό και έχουν περιορισμένους αμυντικούς προπολογισμού. Η Γερμανία μάλιστα έβαλε την ιδέα να δημιουργηθεί αυτό το κόνσεπτ όπου ένα καράτος θα είναι το, το πλαίσιο συνεργασίας το αμυντικό τομέα και θα συνεργάζεται με άλλες χώρες, θα υποβάλει σχέδιο και στο ΝΑΤΟ, αλλά φαντάζομαι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε όλοι, δεν έχουμε όλοι την πολυτέλεια να κάνουμε τα πάντα μεμονωμένα ο καθένας από μόνος του και δεν έχει και νόημα κάτι τέτοιο να κάνουμε ο καθένας ε, το δικό του γιατί οι χώρες έχουν διαφορετικές προτεραιότητες ε, και διαφορετικές ικανότητες αλλά μπορούμε σε μικρότερους σχηματισμούς πολύ πιο ευέλικτους ε, να έχουμε δράσεις που θα τους θέτουμε στη διάθεση, στη διάθεση μετά και το, του συνόλου των συμμάχων. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τζέιμ Απατουράη, τον αναπληρωτή βοηθό Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που ήρθε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και μας ενημέρωσε για την έκβαση της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και φαντάζομαι και στο μέλλον θα σας προσκαλέσουμε. Και ελπίζω να ήταν αμοιβαίως ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψε. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό διάλειμμα και συνεχίζουμε.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 Κυρίε και κύριοι, περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, τα διάφορα. Δεν υπάρχουν διάφορα. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου, 9 το πρωί. Λύεται η συνεδρίαση. Uh, we start in just